Uh, please take a seat, ladies and gentlemen. I'm going to start our afternoon meeting. Να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Βάλτε και τα ακουστικά σας, θα συνεχίσω στα πολωνικά. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην απογευματινή μας συνεδρίαση, η οποία αφορά θέματα αστικού δικαίου. Θα ασχοληθούμε ιδίως με το οικογενειακό δίκαιο. Θα λάβουμε υπόψη βέβαια τις ε, διασυνοριακές του διαστάσεις. Το πρόγραμμα Στοκχόλμης δεν ασχολείται μόνο με την ασφάλεια ή με τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η σύγκρουση των αστικών εθνικών δικαίων δεν μας ενδιαφέρει πολιτικά. όπως μας ενδιαφέρουν τα ποινικά θέματα. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπό την αστική νομοθεσία τα κράτη-μέλη πρέπει άμεσα να εφαρμόσουν στην εσωτερική τους ένομη θάση την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να επηρεάσουμε πολύ αυτή την νομοθεσία. Επίσης, ε, τα θέματα αστικού δικαίου ε, επηρεάζουν την ελευθερία κίνησης των πολιτών, την ελευθερία εγκατάσταση στο κράτος μέλος επιλογής μας. Επηρεάζουν λοιπόν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω ότι με εναρμονισμένα πρότυπα και με την ασφάλεια δικαίου που προσπαθούμε να επιτύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες ρυθμίζονται μέσω του, δουλειά μας. Είμαι επίσης πεπισμένος ότι, ότι αυτά τα θέματα που μόλις ανέφερα θα, μειώ, μειώσουν και τη διάρκεια των διαδικασιών των δικών Και, τα λοιπά και βεβαίως θα μειωθεί και το κόστος που απορρέει από αυτές τις αστικές δίκες. Η δουλειά που κάνουμε για αστικά θέματα, παραδείγματος χάρη ε, ο κανονισμός για το διαζύγιο, ε, ο κανονισμός για τους διεθνείς γάμους, ο κανονισμός για τις κληρονομιές, Όλα αυτά απαιτούν σκληρή και κοπιαστική δουλειά που χρειάζεται χρόνο. Τα συστήματα τα αστικά στα διάφορα κράτη-μέλη, παρότι έχουν τις ίδιες ρίζες και τις ε, ίδιες παραδόσεις, διαφέρουν σημαντικά ως προς τις λεπτομέρειές τους. ούτως ώστε να φτάσουμε σε, στις επιθυμητές λύσεις. Για να φτάσουμε μάλλον σε λύσεις που αποδέχονται όλα τα μέρη, συχνά χρειαζόμαστε μήνες. Δεν είναι εύκολο να φτάσουμε σε συμβασμό. Υπάρχει ας πούμε μεγάλη διαφορά στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες. Και είναι ένας τομέας όπου χρειάζεται μια κάποια εναρμόνιση ορισμένων κανόνων όταν έχουμε να κάνουμε με διασυνοριακές υποθέσεις. Όλα αυτά μας οδήγησαν στην εφαρμογή της αρχής της ενισχυμένης συνεργασίας. Ο κανονισμός για το δικαίωμα επιλογής της δικαιοδοσίας, δηλαδή του δικαστηρίου ουσιαστικά, του αρμόδιου δικαστηρίου σε περιπτώσεις διαζυγίου, ε, είναι η πρώτη απόπειρα για να επιλύσουμε δύσκολες καταστάσεις με διασυνοριακή διάσταση. Εδώ εν προκειμένου παντρεμένα ζευγάρια που προέρχονται από διαφορετικά κράτη-μέλη. Ειδικά όταν τα άτομα, αυτά ή το ένα από τα δύο άτομα δεν μένουν στη χώρα καταγωγής τους. Συχνά τα άτομα αυτά δυσκολεύονται να εξοικειωθούν με τις εγγενείς δυσκολίες του δικαίου της χώρας όπου διαβίουν. Και συχνά μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν και την επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας αυτής. Η επιλογή του δικαίου υπό το οποίο τα ζευγάρια μπορούν να χωρίζουν, να παίρνουν διαζύγιο, είναι τεράστια σημασία λοιπόν. Οι σχετικές δυσκολίες εξάλλου ε, οδήγησαν και σε δραματικές ιστορίες. Έχουμε ακούσει πολλές τέτοιες ε, συναισθηματικά φορτισμένες ιστορίες. Το να θέσουμε λοιπόν ένα κοινό παρανομαστή ελάχιστων κοινών προτύπων, ας πούμε, θα μας εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου. Και είναι πολύ απαραίτητο κατά την άποψή μας κάτι τέτοιο. Τα συστήματα λοιπόν, τα αστικά συστήματα στα κράτη-μέλη διαφέρουν. Ως προς τον ορισμό του γάμου, καταρχήν. Έχουμε τεράστιες ε, διαφορές ήδη στον ορισμό. Και για αυτό το λόγο δεν αποφάσισαν όλα τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη διαδικασία συνεργασίας. 14 κράτη-μέλη αποφάσισαν να το κάνουν μόνο από το 27. Όταν όμως αποδειχθεί η λύση που επιλέξαμε επιτυχής, είμαι σίγουρος ότι και άλλα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν. Στην απογευματινή μας λοιπόν συνάντηση θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν την εναρμόνιση του αστικού δικαίου των κρατών μελών. Θα δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα Πάιν από την Επιτροπή Γιούρε, νομικών υποθέσεων δηλαδή, που είναι η για δύο πολύ σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που αφορούν την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων για το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων και των καταχωρημένων συντρόφων. Εμείς το θέμα αυτό το συζητήσαμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η συνάδελφός μου θα σας πει που φτάσαμε μετά από τις εργασίες της Επιτροπής μας. Να μιλήσω γερμανικά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ψηφίσαμε μόλις σήμερα το πρωί Οπότε τα πράγματα είναι πολύ επίκαιρα και με τους ε, συναδέλφους ψήφισαμε αυτές τις δύο προτάσεις ε, κανονισμού. Δύο αποχές υπήρχαν, ε, μία από έναν Βρετανό, η Βρετανία τους ή άλλους λόγω opt-out δεν συμμετέχει, και άλλη μία γιατί αφορούσε τις καταχωρημένους συντρόφους. Βεβαίω, πολιτικές απόψεις διαφέρουν Έχουμε κράτη-μέλη στα οποία υπάρχουν γάμοι ομοφιλοφίλων, υπάρχουν, υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καν σύμφωνο συμβίωσης. Οπότε έχουμε όλο το φάσμα, τα αποτελέσματα ήταν αυτά τα οποία σας είπα και είχαμε δύο προτάσεις. Η μία αφορούσε συζύγους και καταχωρημένους ε, συντρόφους για να καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις. Γιατί έχουμε και κάποιες καθολικές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, όπου τα σύμφωνα συμβίωση είναι 100% ισότιμα. Το ίδιο ισχύει, όπως είπα, και με τους ε, καταχωρημένους ε, συντρόφους. Στο Βέλγιο, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν ε, κανονικά και γάμοι ομοφιλοφίλων και μη, οπότε, όπως είπα, έπρεπε να διαχωρίσουμε το ζήτημα. Το θέμα λοιπόν είναι το εφαρμοστέο δικαίωμα. Και βεβαίως αυτά είναι τα τελευταία θέματα τα οποία ελπίζω να περάσουν πραγματικά σε αυτή τη θητεία γιατί τότε θα έχουμε κάνει μια μεγάλη επιτυχία και θα έχουμε βοηθήσει τους ε, πολίτες όχι μόνο να συζητάμε συνεχώς τα μεγάλα ζητήματα αλλά να ασχοληθούμε και με τα πρακτικά ε, προβλήματα των πολιτών όταν χωρίζουν ποιος παίρνει τι και τα λοιπά. Επιπλέον, το εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι ενιαίο οπότε δεν θα έχουμε αυτό το οποίο είχαμε μέχρι τώρα ότι ισχύει διαφορετικό δίκαιο για τα ακίνητα από ότι για την κινητή περιουσία. Δεν θα ισχύει πλέον αυτό, δεν θα γίνεται διάκριση μεταξύ κινητών και ακινήτων. Και, όπως προβλέπετε, ε, εξετάζεται κατά κύριο λόγο η τελευταία η πιο πρόσφατη κατοικία και είναι τελείως δευτερεύουσα η υπηκότητα. Βεβαίως ο κύριος Λέχνερ να διευκρινίσουμε τα της ε, κληρονομιάς γιατί πάρα πολλοί θεωρούν ότι αυτό το οποίο κρίνει τα πράγματα είναι η υπηκότητα. Αλλά όπως είπα δεν θα συνεχίσει να ισχύει αυτό, θα εξετάζεται ποια είναι η κοινή κατοικία που είχαν τελευταία αυτοί οι οποίοι χωρίζουν. Και αν έχουν την ίδια επικοότητα ή διαφορετική υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Πολιτικά ήταν το θέμα επίμαχο γιατί ε, είχα προβλέψει την δυνατότητα επιλογής δικαίου και για τους καταχωρημένους συντρόφους. Βεβαίως αυτό για πολλούς ήταν υπερβολικό, αλλά συμφωνήσαμε με τον να μπει στα εκτιμώντας πως μόνο για τους σκοπούς ε, του κανονισμού αυτού η καταχωρημένη σύντροφοι είναι κάτι το διαφορετικό από παντρεμένους. Βεβαίως ήταν μεγάλες οι πολιτικές συζητήσεις γιατί εγώ είχα παγιδευτεί μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχει πλήρης ισοτιμία και των κρατών μελών όπου υπάρχουν σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Να, να δώσω ένα παράδειγμα στο μέλλον. Αν δύο Γερμανοί έχουν ε, μια, ένα σύμφωνο συμβίωσης Γερμανία και πάνε στην Πολωνία για να εργαστούν. Η Πολωνία δεν αναγνωρίζει ε, το σύμφωνο αυτό συμβίωσης, οπότε δεν θα μπορέσουν να χωρίσουν εκεί γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί, κανένα δικαστήριο σε κράτος μέλος δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να αποφασίσει για κάτι τέτοιο, αν δεν υφίσταται καν ε, τέτοιος θεσμός. Γιατί υπήρχε ο φόβος των κρατών μελών πως οι πολίτες τους θα χρησιμοποιούν το δίκαιο ενός άλλου κράτους μέλους για να εκμεταλλευτούν τον θεσμό του Συμφώνου Συμβίωσης πριν εισαχθεί σε άλλες χώρες. Οπότε αποκλείσαμε. Κανένα κράτος δεν θα αναγκαστεί να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο δικό του δίκαιο. Ψηφίσαμε σήμερα το πρωί. Σε δύο μήνες θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Στο Συμβούλιο τα πράγματα είναι ως εξής. Ε, δεν είναι στη διαδικασία της συναπόφασης, είναι απλά μία διαδικασία διαβούλευσης. αλλά βέβαια ε, θα μπορούσαμε να έχουμε τη διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας, ε, όπως είπε και ο κ. Σφίφκα, αλλά βεβαίως αυτό δεν έγινε λόγω της ε, Σουηδίας, γιατί όπως είπα τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν πλήρη ισοτιμία έχουν το πρόβλημα με τις χώρες που δεν υπάρχει πλήρης ισοτιμία. Αλλά στο Συμβούλιο συμβαίνει το εξής. Όλα τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν ίση αντιμετώπιση και με τις δύο μορφές. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγα κράτη-μέλη που είναι κατά της δυνατότητας επιλογής δικαίου για καταχωρημένους συντρόφους. Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία, κάπως έτσι κέντρο ευρωπαϊκές ε, χώρες αλλά ελπίζουμε πως θα καταλήξουμε σε κάποια απόφαση γιατί τελικά τα πράγματα προς μία κατεύθυνση πηγαίνουν η αλλαγή της νομοθεσίας στη Γαλλία νομίζω πως ήταν μεγάλη όθηση για τις προτάσεις αυτές κανονισμού με βοήθησε μέρα στη δουλειά μου για ό,τι άλλο θέλετε είμαι στην διάθεσή σας είναι πολύ τεχνικό το ζήτημα. Είχαμε και κάποια ζητήματα με την Γαλλία όσον αφορά το τι γίνεται στη Γαλλία με κοινά αποκτήματα αλλά και κάποια επιδόματα στην Γερμανία που το άφησαμε εκτός γιατί ήταν ε, εκτός Αυτά λοιπόν για τίποτα άλλο στην διάθεσή σα. Αλεξάνδρα, Ευχαριστώ. Αλεξάνδρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω μια διαδικασία που είναι γνωστή ήδη σε εσά. Για το πώς παίρνουμε το λόγο στη συζήτηση. θα μπορέσετε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας τα έντυπα που σας έχουμε δώσει. Θα τα συμπληρώσετε, θα τα μαζέψουμε και θα τα κοιτάξουμε. Ούτω ώστε να μπορέσετε να πάρετε το λόγο στη συζήτηση αργότερα. Τώρα θα δώσω το λόγο σε έναν πρώην Ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Κέρτ Λέχνερ, ήταν ευρωβουλευτή μέχρι πριν από λίγους μήνες. Και μάλιστα στο τέλος, κατά το τέλος της θητείας του ήταν και εισηγητής σε μια έκθεση που αφορούσε διασυνοριακές κληρονομιάς. Η δουλειά του ήταν καταπληκτική. Χρειάστηκε να λάβει υπόψη καταρχάς τις διαφορετικές παραδόσεις στο διαφορά το κληρονομικό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Ο Κούρτ λοιπόν θα σε μιλήσει για την εμπειρία του, θα σα δώσει διάφορες λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή που, είχε, που διαπραγματευθήκαμε. Ευχαριστώ Ταντέους. Έχω τώρα που έχω αποσυρθεί λίγο περισσότερο χρόνο για να ασχοληθώ με ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούσαν και ελπίζω όπως είπα να οδηγηθούμε σε επιτυχία αλλά θα ήθελα να πω πως η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με πριν 10-12 χρόνια όταν πρώτο ήρθα στο Κοινοβούλιο τότε είχα ασχοληθεί με το δίκαιο της χρεοκοπίας και Είχαμε κάνει πολλές προτάσεις, τότε δεν, δεν ενδιαφέρανε καθόλου το Συμβούλιο. Βεβαίως, εντωμεταξύ έχει αλλάξει η κατάσταση. Τώρα να πω για τους συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν πως είναι ενδιαφέρον πως πριν από λίγες εβδομάδες, μήνες υπογράφτηκε μια γαλλογερμανική συμφωνία ακριβώς για το θέμα της ε, κληρονομικής διαδοχής, ε, ουσιαστικό δίκαιο, κάτι το οποίο δείχνει πως ε, υπάρχει κάποια σύγκληση στην Ευρώπη τώρα για τον κανονισμό αυτόν. Δεν ήταν το πρώτο θέμα στο οποίο ήμουν ο εισηγητής και ήμουν στις διαπραγματεύσεις. χρειάζεται λίγος μαζοχισμός για αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά περιέργως ήταν η τελευταία διαπραγμάτευση και η δυσκολότερη, αλλά και η πιο επιτυχής ε, ε, περιέργως ε, στο τέλος της βουλευτικής μου Και ήταν ευχάριστη γιατί το κλίμα των διαπραγματεύσεων και στο Κοινοβούλιο, αλλά και με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό και παρόλες τις διαφορές απόψεων ε, και αποκλήσεις ε, συνολικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να αναφέρω εδώ πέρα και την Κομισιόν από την οποία ίσως θα περίμενε κανείς ε, να υπερασπίζει την πρότασή της σε όλες τις λεπτομέρειες. Αντιθέτως η Κομισιόν ευχαρίστως προσέφερε τις υπηρεσίες της που ήταν πάρα πολύ υψηλού επίπεδου για να βελτιώσει τις δικές μας ε, προτάσεις. Και όλοι οι εκπρόσωποι της ε, Κομισιόν, τέσσερα άτομα με τα οποία ε, συνεργάστηκα και ήταν ικανότατοι και ήταν γυναίκες επίσης, κάτι το οποίο ίσως βοήθησε το κλίμα. Πρέπει επίσης να πούμε πως υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στο θέμα αυτό. Πρέπει να πω και στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κινείται στην κατεύθυνση κυβέρνησης αντιπολίτευσης όπως τα Εθνικά Κοινοβούλια. Παρ' αυτά οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις παίζουν μεγάλο ρόλο και θεωρώ πως ε, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται πάντα με μια συνένεση στα πάντα και δεν διακρίνει καμία διαφορά ο πολίτης. Ε, πρέπει να υπάρχει και κάποια διαφορά. Αλλά στο θέμα αυτό που είναι θέμα ιδιωτικού δικαίου οι πολιτικές κατευθύνσεις δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, ήταν περισσότερο θέμα εθνικών παραδόσεων που ήταν ε, σημαντικές ε, και αντικρουόμενες και ήταν ε, τεχνικά δύσκολο το ζήτημα. Και εκεί πέρα, όπως σας είπα, αφήσαμε κατά μέρος το ουσιαστικό δίκαιο, καθώς εκεί πέρα είμαι κάπως επιφυλακτικός όσον αφορά την προσέγγιση. Αλλά παρόλα αυτά το ανέφερε και ο Τοντέρος Βιφκά, πως καμιά φορά όταν τεχνικά τα πράγματα κυλάνε πιο γρήγορα αλλά στην περίπτωσή μας υπήρχαν παραδόσεις αιώνων των κρατών μελών που έπρεπε να αλλάξουν πολλά κρατημέλη έχουν ως αφετηρία και βασικό κριτήριο την υπηκότητα αλλά τον τόπο κατοικίας. Δικαίωμα επιλογής δεν υπήρχε σε κανένα κράτος μέλος. Ε, μιλάμε δηλαδή για σοβαρότατες αλλαγές ε, που είχαν ε, και επιδράσεις όπως είπα στο ουσιαστικό δίκαιο και γι' αυτό όπως είπα υπήρξε μια προσέγγιση για να ακολουθήσουμε έτσι μια συνενετική διαδικασία με τα κράτη-μέλη και με τη βοήθεια της Κομισιόν. ανοίξαμε όλα τα ζητήματα, όλα τα προβλήματα τα συζητήσαμε, δεν αγνοήσαμε τίποτα. Ζητήματα διαδικαστικά, δικαιοδοσίας, υπάρχουν πάρα πολλά γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι διαφορές ε, των κρατών μελών και όλα αυτά τα συζητήσαμε άνοιχτα και είχαμε έναν συνεχή διάλογο και εδώ στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό, αλλά και με τους εθνικούς συναδέλφους. Είχαμε κάποιες συναντήσεις με την Κομισιόν, με το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη και με εμπειρογνώμονες, με μελέτες, ακροάσεις ε, και με την κοινωνία των πολιτών, δικηγόρους, δικαστές, ενώσεις ε, συμβολεογράφων και όπως είπε και ο κύριος Σοτσφίφκα, χρειάζεται χρόνος και υπομονή. Δεν έχει νόημα ένα τόσο ευαίσθητο θέμα να το προσεγγίζει κανείς με τρόπο χοντροειδή. Να δώσω ένα παράδειγμα, ένα υποπροϊόν σχεδόν της όλης διαδικασίας, ε, το οποίο δεν είχα σκεφτεί. Είχαμε συζητήσει πάρα, πολύ, πάρα πολλές φορές με την κυρία Φαντεκέρ Χόφε του Κομισιόν, αλλά και το ζήτημα της ε, διασυνοριακής αναγνώρισης ε, πιστοποιητικών με το Συμβούλιο και πραγματικά καταλήξαμε στην ε, πρώτη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η ισχύς ε, ειδικά των ε, συμβολιογραφικών πράξεων επεκτάθηκε διασυνοριακά. Και είναι πραγματικά, όπως σας είπα, ένα από τα προϊόντα αυτής της ε, διαδικασίας. Είχαμε συνεχείς συζητήσεις, συναντήσεις με όλους ε, τους συμμετέχοντες και υπήρχε μεγάλη διάθεση συνεργασίας. Και η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα ήταν πως είχα την εντύπωση πως όλοι ήθελαν την επιτυχία. Δεν ε, μπλοκάριζε κανείς τίποτα. Υπήρχαν επιφυλάξεις, τα κράτη-μέλη είχαν τις ιδιαιτερότητές τους για τις οποίες πάλεψαν, αλλά και στο Κοινοβούλιο και οι βουλευτές το ίδιο, αλλά κανένας δεν ε, μπλόκαρε τη διαδικασία. Και, σας είπα, είδαν όλοι το σύνολο και όχι μόνο τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Κανείς δεν μπορεί να πει λοιπόν πως ε, εμείς κερδίσαμε, περάσαμε το δικό μας. Είναι όλα αυτά που σας είπα, είναι καινούργια για όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι άλλο για την αρχή της πλειοψηφίας. Στην όλη διαδικασία της ε, συναπόφασης, η όλη διαδικασία της συναπόφασης έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία. Και είναι κρίμα το ότι δεν υπήρχε εδώ πέρα ε, η αρχή αυτή. Γιατί, κοιτάξτε, ε, η απόφαση του Κοινοβουλίου επιδρά και στο Συμβούλιο. Όταν ε, μια επιτροπή του Κοινοβουλίου λαμβάνει μια απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία, παρακινείται και το Συμβούλιο να ακολουθήσει. Και βεβαίως ε, όταν, ε, όπως συμβαίνει και γενικότερα και στον ιδιωτικό βίο, σε αυτές τις περιπτώσεις ε, υπάρχει κάποια συνένεση. Και αντιστρόφως βεβαίως, όταν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις ε, πάλι γίνονται συμβιβασμοί γιατί αλλιώς άμα είναι οι αποφάσεις ομόφωνες δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Οπότε συνολικά θα έλεγα καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα και όλα αυτά συνεισέφεραν σε ένα σε συνετικό αποτέλεσμα. Να αναφέρω κάτι άλλο, ένα άλλο παράδειγμα. Ε, σημαντικό σημαντικό θέμα του, που απασχόλησε το Κοινοβούλιο ήταν η δυνατότητα να επιλεγεί το δίκαιο σε χώρες όπως η Πολωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, όπου έπαιζε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η υπηκότητα. Γιατί βεβαίως ε, έγραφε ο κόσμος ε, μια διαθήκη και ε, ήταν εννοείτο ότι θα ίσχυε το δίκαιο της ε, υπηκότητάς του. Το ξεκαθαρίσαμε όμως ότι πρέπει πλέον να δηλώνεται ρητός, όχι απλά να εννοείται, το ότι θα ισχύει το άλλο δίκαιο, το, το χύψη δίκαιο. Και το αιτιολογήσαμε με τη λογική και των υπολείπων ε, συμβάσεων όταν γίνονται συμβάσεις ε, μεταξύ δύο μερών ε, γιατί βεβαίως πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ δύο μερών μπορεί να ερμηνευτεί η σύμβαση αλλά βεβαίως η Διαθήκη δεν είναι πια αντικείμενο ερμηνείας οπότε υπό την ηγεσία θα έλεγα της Ανίας καταλήξαμε και εκεί πέρα σε ένα αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω κάτι τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ε, επέλεξαν να μην ε, ενταχθούν. Και άλλη μια διαφορετική κατάσταση υπάρχει στην Δανία. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί τα προβλήματα που είχε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σοβαρά και κατανοητά, δεν το συζητάει κανείς αυτό. Αλλά το Ενωμένο Βασίλειο βεβαίως συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, επηρέασε τις διαπραγματεύσεις και ψήφιζαν οι βουλευτές του, οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο. Και βεβαίως δεν είχαν να σκεφτούν το τι θα γίνει στο τέλος, να ψηφίσουν για συμβιβασμό και τα λοιπά, γιατί τους ήταν αδιάφορο το ζήτημα. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα λοιπόν για εμάς ε, και για τους υπολείπους ε, συναδέλφους. Οπότε, εντάξει, μία φορά να γίνει, αλλά το αν είναι κανόνας ε, αυτή η πρακτική δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν θέλω να απευθύνω κάποια μομφή, ήταν σοβαρό το πρόβλημα του Ηνωμένου Βασιλείου, πράγματι εντάξει και η Γερμανία είχε. Εντάξει, ίσως να μην ήταν τόσο, τόσο σημαντικό. Λοιπόν, η όλη διαδικασία, η συζήτηση κράτησε 1,5 χρόνο. Όπως σας είπα ήταν προσανατολισμένη στην ουσία, καταλήξαμε νομίζω σε ένα καλό αποτέλεσμα, καλύτερο από την πρόταση της Κομισιόν και Μάλιστα, χάρη στην ε, συνεργασία και τη βούληση για συνεργασία όλων των συμμετεχόντων της ε, Κομισιόν ε, και του Συμβουλίου σε όλες τις προεδρίες νομίζω άξιζε και ο κόπος και ο χρόνος που αφιέρωσαμε. Ευχαριστώ. Κουρτ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Όντως, Πρόκειται για ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει κατά τι εργασίε τη Νομική Επιτροπή και ανακύπτουν ε, ουσιαστικά καθημερινά. Θα πρέπει κανεί να ξεχωρίσει τι θα πρέπει να εναρμενιστεί και τι όχι. Είναι αλλιώ η καθηγορία γιατί θυμάμαι ότι είχα πάει σε κάποιο συνέδριο συμβολιογράφων στην Αυστρία για θέματα αστικού κώδικα. Και μα ρωτάγανε γιατί θέλει το Κοινοβούλιο εναρμόνιση στο οικογενειακό δίκαιο. Όχι, δεν θέλουμε έναν ε, ευρωπαϊκό αστικό κώδικα. Όμως υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα θέματα όπου αν κανεί λάβει υπόψη την ε, κινητικότητα των Ευρωπαίων και τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της ε, ε, της ε, κινητικότητας χρειάζεται να υπάρξει αυτή η ενερμόνιση. Φυσικά με το ζόρι τίποτα δεν γίνεται. Με το ζόρι τίποτα θέλουμε να επιβάλλουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε για τις προθέσεις μας. Προσπαθούμε να εξεύρουμε έναν συμβασμό και να προκύψουν λύσεις που να ικανοποιούν τους πάντες πάρα πολύ συχνά στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχουμε συζητήσεις που αφορούν την επιλογή της πιο κατάλληλης νομικής βάσης. Με πολύ σημαντικό κάθε φορά ποιο άρθρο της συνθήκης θα επιλέγεται ως νομική βάση για αληθεί κάποιο νομικό θέμα. πρόκειται για περίπλοκη συζήτηση, ξέρετε. Γιατί κάθε φορά έχει κανείς να αντιμετωπίσει διαφορετικές νομικές παραδόσεις του κάθε κράτους. Ανάλογα με το ποιοι είναι οι μπλεκόμενοι δηλαδή βουλευτές. Η συγγήτρια είναι η Οντ Φιωρίνη από το Πανεπιστήμιο του Νταντή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. To give me the opportunity to participate in this exchange of views today. Um, as we've already heard, um... Όπως ε, ήδη ακούσατε λέει κυρία Φιωρίνη, η εξέλιξη του οικογενειακού δικαίου είναι θεαματική και συνεχίζει. Τα τελευταία 12-13 χρόνια είχαμε μόνο σαν κοινέ διατάξει μόνο τα της διατροφή αλλά τώρα ε, έχουμε ένα σωρό διατάξεις ε, που αρπούμε την Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Δικαίου. Ακούσατε από τις προηγούμενες και αυτή η εξέλιξη στο Οικογενειακό Δίκαιο ήταν ε, βραδύτερη, ήταν πιο δύσκολη από όσο σε άλλα ζητήματα εμπορικού δικαίου ή άλλα ζητήματα αστικού δικαίου. Χρειάζεται ειδική νομοθετική διαδικασία. Σύμφωνα με τη συνθήκη γίνεται μια διάκριση. Χρειάζεται ειδική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 3. Πρώτο εδάφιο. Οπότε και έτσι έχουμε κάποιες ε, διατάξεις είτε για όλα τα κρατημέλη ή για συγκεκριμένα σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας της ενισχυμένης εργασίας. Όμως, κάτι εξαίρεση. Εάν χρησιμοποιήσουμε την ε, μεταβατική ρήτρα, μπορούμε να έχουμε την συνήθεια νομοθετική διαδικασία και για ζητήματα κοινωνικού δικαίου. Και εξηγούμε. Η μεταβατική ρήτρα σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι ελαφρώς διαφορετικό από την ρήτρα που χρησιμοποιείται στα ζητήματα ενισχυμένης συνεργασίας. Χρειάζεται διαβούλευση για τα ζητήματα κοινωνικού δικαίου και επίσης χρειάζεται ομοφωνία. Όλοι γνωρίζετε γιατί υπάρχει αυτή η ειδική ρύθμιση και μεταχείριση για τα ζητήματα του κοινωνικού δικαίου. Γιατί είναι ζητήματα ιδιαίτερα ευαίσθητα, ιδιαίτερα δύσκολα ε, και είναι επίσης και βαθιά ριζωμένες παραδόσεις και κουλτούρα του κάθε λαού. Όμως, εδώ υπάρχει κάποιο παράδοξο κατά κάποιο τρόπο. Αυτή η ειδική ρύθμιση και μεταχείριση έχει ένα τίμημα. Θα συμφωνείτε ότι το πυριακό δικαίωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαίο. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ζήτημα όπου οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων δεν έχουν το ίδιο πλήρη αρμοδιότητα όπως στην περίπτωση της συναποφάσεως. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινωνικό δίκαιο. Και το ότι απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο, αυτό οδήγησε στην βραδία εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου. Μπορούν επίσης να προβαλούν βέτο ε, κάποια κράτη για να προστατεύσουν κάποιο εθνικό συμφέρον, εθνική πολιτική. Ή πολλές φορές θεσπίζεται ένας κανόνας, αλλά με αντάλλαγμα κάποιο είδους ε, ε, συμβιβασμό επώδυνο που μπορεί να απονευρώσει τους σκοπούς του θεσπιστέντος μέτρου νομοθετήματος. Επομένως θα πρέπει ή όχι να χρησιμοποιείται η μεταβατική ρήτρα. Σε αυτή την περίπτωση η συνήθις διαδικασία οδηγεί σε ευρύτερο διοργανικό διάλογο και κατά πλειοψηφία ψήφο στο Συμβούλιο. άποψη λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τα μεταβατική γιατί είπαμε ότι έτσι αλλοιώνεται η ρύθμιση σε τεμινοτομία τόσο λεπτό. Έχουμε άλλωστε και το 67 της ε, Συνθήκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ορίζεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Με σεβασμό στα δικαιώματα και στις διαφορετικές νομικές παραδόσεις των κρατών μελών. Πάραθα να μην υπερβάλλουμε όσον αφορά τη δυσκολία αυτού του προβλήματος. Γιατί δεν είναι και τόσο μεγάλη η, η παραβίαση της ε, εθνικής ακυριότητας από την χρήση της μεταβατικής ρήτρας. Μια που και η επιτελετική ρήτρα απαιτεί ομοφωνία στο Συμβουλίο. Επίσης χρειάζεται και επικύρωση της σχετική απόφαση από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όμως, έχουμε την εξαίρεση από αυτή τη ρύθμιση, δηλαδή την επικύρωση από την Ευρωκοινοβούλια, εάν ισχύει το άρθρο 333 παραγράφος 2. Τώρα, να δούμε τώρα, αν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα οικογενειακού δικαίου, στα οποία δεν συνιστάται η χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Πάντω η απάντηση που θα δώσουμε σε αυτό το ερώτημα δεν εξαρτάται από το συγκεκριμένο ζήτημα οικονομικού δικαίου, αλλά κυρίω όσον αφορά το ζήτημα ουσία και όσον αφορά το, το πεδίο εφαρμογή, το εύρο, το ελληνικέ του προτείνουμε νομοθετήματο. Γιατί έχουμε κάποιες, ε, ε τομείς του δικαίου, δηλαδή ε, έχουμε κάποια σημεία που συναντά το κοινωνικό δίκαιο με το ενοχικό δίκαιο ή το εμπράγματο δίκαιο. Α, και πριν που μιλούσαμε για το κληρονομικό δίκαιο. Και έχουμε αυτές τις, ε, επομένως, τις, ε, τα, τα μεικτά νομικά ζητήματα, στα οποία δεν προσφέρεται τόσο πολύ η χρήση της μεταβατικής ρήτρας. Οπότε και αυτά τα νομικά ζητήματα είναι το ίδιο σημαντικά όπω, το ποινικό δίκαιο. Επομένω τελικά είναι θέμα περιεχομένου. Επίσης, έχει διατυπωθεί άποψη ότι η χρήση της μεταβατικής ρήτρας προσφέρεται όποτε τα μέτρα αφορούν υπάρχουσα εναρμόνιση, ας πούμε μέσω απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή επειδή προϋπήρχε μια διεθνή σύμβαση την οποία τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα συμπληρώνουν ή παγιώνουν. Επίσης, προσφέρεται η μεταβατική ρήτρα εάν έχουμε ένα μέτρο το οποίο ενσωματώνει κάποιες αρχές οι οποίες είναι αποδεκτές από όλα τα κρατημέλη. Πάντως ενδεχομένω να μην είναι δυνατόν να υπάρχει συμφωνία από αυτού, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια άλλη δυνατότητα. Έχουμε τις διατάξεις της ε, ενισχυμένης συνεργασίας. Προβλέπουν οι συνθήκες τέλο πάντων αυτήν την περίπτωση υπό κάποιες προϋποθέσεις διαδικαστικές και ουσιαστικές. Αλλά στο άρθρο 20 πάντως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές προϋποθέσεις για την ενισχυμένη συνεργασία. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως τελευταία λύση, έσχατη λύση. Και επίσης ότι θα πρέπει αυτό να προωθεί, να προαγάγει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα πει τώρα έσχατη λύση, τι θα πει έσχατη καταφυγή. Κανείς δεν ξέρει γιατί η συνθήκη δεν δίνει έναν ορισμό. Το μόνο το οποίο αναφέρω στις συνθήκες είναι ότι όταν οι στόχοι του μέτρου δεν μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε ένα λογικό, εύλογο διάστημα από το σύνολο της Ένωσης. Να, αυτό με κάπως μας βοηθάει λίγο. This, um, um, which has um, given a little more precision on last resort and um, uh, specified at last. Θα πρέπει βέβαια να περιχαρακωθεί αυτός ο ορισμός με κάποια περισσότερη ακρίβεια. Και να δούμε κατά πόσον έτσι μπορεί να εφαρμόζεται αυτή η διάταξη ή θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Πάντως, είναι θέμα του ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος στον οποίο κατατείνει ένα νομοθέτημα. Μήπως μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους το ίδιο δόκιμος. Άρα, τι θα γίνει αν έχουμε διαπραγματεύσει για ένα ε, μέτρο που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι διαπραγματεύσει αυτέ πέσουν στο κενό. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, μήπω τότε θα πρέπει να έχουμε την σημαίνει συνεργασία. Να και να θεωρείται τότε ότι συντρέχει περίπτωση επομένω σε τη καταφυγή, σε τη λύσεω. Πάντω αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το κοινωνικό δίκαιο. Το θέμα είναι αν θα πρέπει να υπάρχει ή όχι ενισχυμένη συνεργασία. Αν θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος για, τους, ε, για κάποιους για όλους τους Ευρωπαίους. Δεν μπορούμε να δώσουμε ορμένως απάντηση, απλώς θα να διαφωτίσουμε την κατάσταση. Πάντως εύκολα μπορεί κανείς να πέσει σε σύγχυση αν δεν ξεκαθαριστεί ότι υπάρχουν δύο είδη ε, ή στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 20 των συνθήκων. Στόχοι συγκεκριμένου μέτρου ή νομοθετήματος και στόχοι της Ένωσης. As was said um, previously, of course, enhanced cooperation. Um, um, Οπότε ε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί να είναι καταλήτης και για άλλες χώρες που θα έρθουν να ενωθούν, να συμμετάσχουν στην συνεργασία με τα συνεργαζόμενα κράτη-μέλη. Επίσης, είναι δυνατόν αυτή η ενσυμμένη συνεργασία να αποτελεί την ε, αφορμή να ξεκινήσει μία ευρύτερη μεταβλητή γεωμετρία. Οπότε, βλέπουμε ότι δεν είναι πανάκια αυτή η μέθοδος, διότι το ευρωπαϊκό Γενικό δίκαιο είναι αστομίας όπου δεν έχουν στενά εδαφική εφαρμογή τα θεσπιζόμενα νομοθετήματα. Επίσης, τελικά έτσι πλήσεται και η ασφάλεια δικαίου. Όμως, η ασφάλεια δικαίου είναι ουσιαστικό συστατικό και προαπαιτούμενο για τον χώρο δικαιοσύνης, αυθεντικής δικαιοσύνης που αποτελεί στόχο τη Ένωση. Επομένως, η ενισχυμένη συνεργασία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι δόκιμο να χρησιμοποιείται μόνο κάτι εξαίρεση, σαν τελευταία λύση, έσχατη καταφυγή. Και συμφωνώ με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έκρινε το δικαστήριο ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης δεν μπορεί να προστατευτεί εάν οι διαπραγματεύσει, δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποιο είδου περίπτωση ε, της εργασίας και σε κάποιο είδου συμβασμό, οπότε χρειάζεται να υπάρξει ε, κάποιο είδου νομοθεσία που να εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φιωρίνη για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά την νομική βάση που χρησιμοποιούμε στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Ιδανικά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εντός του χρονικού πλαισίου δεν έχουμε πρόβλημα χρόνου. Έχω δύο μιλητέ στον κατάλογο που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Όσοι δεν έχουν δηλώσει γραπτό ενδιαφέρον, μπορούν παρόλα αυτά να εκφράσουν ενδιαφέρον προφορικά. Ο κύριος ε, Φαμιλιέτη από την Ιταλία τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Η δικαστική συνεργασία για αστικά θέματα είναι ένα από τα πιο προκεχωρημένα σημεία ε, σύγκληση των εθνικών νομοθεσιών. Η συνθήκη της Λισαβόνας καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να ε, υλοποιήσουμε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η διευκόλυνση και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική γιατί ε, πολλοί δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα ε, σχετικό πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού, των δικαστών δηλαδή. Τα, οι πρόοδοι που, σημειω, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μας δίνουν πάρα πολλές ελπίδες για την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει έναν αποφασιστικό ρόλο και σε αυτόν τον τομέα, όπως έχει παίξει και σε άλλους τομείς, για το καλό της ε, ανάπτυξης μεταξύ άλλων. Ε, όλη η νομοθεσία που έχει προωθηθεί για την, τον ανταγωνισμό και την ενιαία αγορά ε, μειώνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και δίνει περισσότερες εγγυήσεις ε, σε πολλούς πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο επίσης μειώνεται ο το κόστος και μειώνται και οι προθεσμίες για την έκδοση και εκτέλεση των αποφάσεων. Μην ξεχνάτε ότι στην Ιταλία, ας πούμε, ο χρόνος εκτέλεσης των αποφάσεων και έκδοση των αποφάσεων είναι πολύ μεγάλος. Έτσι λοιπόν, ο καθένας θα έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην προστασία των δικαιωμάτων του και σε πρόσβαση σε καταρτισμένους νομομαθείς. Τα εργαλεία που προωθούμε στον αστικό τομέα είναι πολύ σημαντικό και για την έννοια της ηθαγένειας. Πρέπει όμως να πάρουν απτή μορφή αυτά τα εργαλεία για να μπορεί να υποφεληθεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Επίσης, υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία απαραίτητα στον τομέα του αστικού δικαίου. Έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα, έχουν να κάνουν με την πολιτική και συνταγματική δομή του κάθε κρατούς μέλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σεβαστεί ε, με βάση το άρθρο της ε, Συνθήκης 4 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ταυτότητα των κρατών μελών. Η Αλεσάνδρα Τέιν μίλησε πολύ σωστά για την ανάγκη να παντρέψουμε αυτό το ταχύ τρένο των μεταρρυθμίσεων της Ευρώπης με τον το ρυθμό με τον οποίο λειτουργούν, κινούνται, τρέχουν ή υπερπατούν απλώς τα κράτη-μέλη. Η υπερπατουν απλω τα Βουλή εξέτασε κάποιες από τις πιο πρόσφατες και σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της ε, συνεργασίας για αστικά θέματα ε, και την πρόταση κανονισμού για τις κληρονομιές. Επίσης, ε, ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου. Η άποψη της Βουλής μας είναι ότι δεν θα αντιταχθούμε στην ε, υιοθέτηση αυτών των προτάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η Ιταλική Βουλή είπε ότι δεν πρέπει να, να ζημιώσουμε τα... τις ιδιαίτερες προστασίες μεταξύ των οποίων κάποιες... όπου κάποιες ε, εθνικές νομοθεσίες επιφυλάσσουν σε ορισμένους πολίτες, ε, μεταξύ των οποίων και το Ιταλικό δίκαιο. Φερρυπίν τα δικαιώματα των κληρονόμων. Θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες προοδευτικά να συγκλίνουν μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ όταν ε, υπάρχουν ε, εδώ ειδικέ ρυθμίσεις εθνικών ένομων τάξεων. Θα πρέπει πάντα η δικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διαφανής ούτω ώστε να φτάσουμε σε τεκμηριωμένες αποφάσεις ε, που θα τις συμμερίζεται μια πλατιά πλειοψηφία κρατών μελών. Ε, με αυτόν τον τρόπο, αν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζουμε και τις ε, αντιευρωπαϊκές τάσεις και εξάρσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαμιλιέτη. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Αλεξάνδερ Πότσεϊ από την Πολωνία. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μιλήσω λίγο στα γαλλικά στην αρχή για να τιμήσω την πόλη στην οποία βρισκόμαστε και όλους τους γαλλόφωνους συναδέλφους. Αλλά μια και ο πρόεδρος είναι Πολωνός, καλό είναι να συνεχίσω στα πολωνικά. Ε, Καταρχήν. Γιατί. Άκουσα τα όσα είπε η κυρία Τάιν και θα ήθελα να ανταπαντήσω τα εξή. Στην Πολωνία ε, ασχολούμαστε ε, με τους καταχωρημένους συντρόφους. Τους, τους λεγόμενους συντρόφους που έχουν συνάψει τα ΠΑΞ, όπως λέμε στη Γαλλία. Η πρώτη απόπειρα απέτυχε. Εγώ και το πολιτικό μου κόμμα, η αστική πλατφόρμα, είναι υπέρ αυτών των καταχωρημένων ε, σχέσεων. Όμως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε οποιαδήποτε λύση σε αυτόν τον τομέα, σε οποιαδήποτε χώρα. Και εδώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Ιταλός συνάδελφος. Το όλο θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ αμφιλεγόμενο. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε σε διεθνές επίπεδο. έχουν γίνει τις προσπάθειες, αλλά έχουν αποτύχει. Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν ε, μείζονες διαφορές. Οι κουλτούρες μας είναι διαφορετικές, οι νομικές μας παραδόσεις είναι διαφορετικές και οποιασδήποτε προσπάθειες εναρμόνισης είναι εξορισμού επικίνδυνες. Να πω δύο λόγια για τη Γαλλία. Η Γαλλία επέτρεψε το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό δίνει πολύ τροφή προς προβληματισμό σε όλους μας. Έγιναν απίστευτες διαδηλώσεις στη Γαλλία, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους να διαδηλώσει την αντίθεσή του και αυτό δείχνει πόσο λεπτό και ευαίσθητο είναι το όλο θέμα. Αλλά σε επανέλθω στην Πολωνία. Αν δεχτούμε τις, καταχωρισμέ... τις καταχωρημένες σχέσεις, όταν οι ομοφιλόφιλοι ζητούν γάμο κανονικό, αυτό θα είναι ε, επιχείρημα εναντίον της αναγνώρισης οποιασδήποτε επίσημη σχέσης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ορισμένοι λένε ότι αν δώσουμε το πράσινο χώρο στις καταχωρημένες σχέσεις, αυτό θα ανοίξει το δρόμο στους γάμους. αυτό όμως είναι απαράδεκτο για την Πολωνία και άλλες χώρες. Δυστυχώς τέτοιου τύπου επιχειρήματα ακούγονται σε αυτές τις συζητήσεις και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, να μην τα ξεχνάμε. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο σε αυτά που είπε η κυρία Τάιν. Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο. Η Πολωνία θέλει να έχουμε αντικειμενικούς διασυνοριακούς κανόνες. Είναι προς το συμφέρον μας. Θέλουμε οπωσδήποτε τους κανόνες. Δυστυχώς η εμπειρία μας μέχρι τούδε ήταν αρνητική. Μιλάω για δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά από διεθνείς γάμους. Δηλαδή, ας πούμε, ο ένας σύζυγος είναι Πολωνός και ο άλλος ξένος. Ήταν πολύ πικρή εμπειρία. Από ό,τι φαίνεται, εμείς Πολωνία έχουμε την τάση να μεταναστεύουμε. Στην Γαλλία, στο Μένο Βασίλειο και στις σκανδιναβικές χώρες. Αυτά τα λέω από την ε, εμπειρία μου και μιλάω ως δικηγόρος που εξειδικεύεται στο οικογενειακό δίκαιο. Σε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν, σε όλες, σχεδόν όλες τις ε, διασυνοριακές ε, περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν ο Πολωνός σύντροφος ή σύζυγος ήταν Πολο... ήταν άντρας ή γυναίκα, η κυδαιμονία, σχεδόν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κυδαιμονία του παιδιού δόθηκε στη χώρα όπου γεννήθηκε το παιδί. Στην Πολωνία όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε εμά το 90% των περιπτώσεων τα παιδιά μετά το διαζύγιο τα παίρνει η μητέρα. Η μητέρα έχει την κυδαιμονία. Ενώ όπως σας είπα σε αυτές τις υποθέσεις το παιδί πήγαινε στο γονιό της χώρας όπου γεννήθηκε. Αν θέλουμε τώρα να ρυθμίζουμε τα θέματα αυτά με βάση κειμένικά κριτήρια, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την ευημερία του παιδιού. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο. Η ευημερία του παιδιού και όχι η χώρα του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται τις υπόθεσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό θέμα. Επίσης, να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα άλλο θέμα που αφορά όχι μόνο Πολωνούς, αλλά και άλλους υπήκους και μάλιστα και υπηκούς τρίτων χωρών. Την Νορβηγία, τη Σουηδία, λέει ο μιλητής, και τη Γερμανία. Έχουμε αυτό το τρίγωνο χώρων. Από ό,τι φαίνεται, πολύ ε, εύκολα τα παιδιά μεταναστών, Πολωνών ή και άλλων χωρών, συχνά τα δίνουν στην κυδαιμονία άλλων ανθρώπων. Αν κατά την άποψη των αρχών ο Πολωνός γονιός έχει κάνει κάτι λάθος. Η παραμικρή, το παραμικρό αδίκημα οδηγείται στο να δοθεί το παιδί σε μία ανάδοχη οικογένεια και όχι στον πολωνό γονιό. Αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να ρυθμιστεί. Επίσης, ε, θα, εμείς θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε τη δουλειά που γίνεται σε αυτά τα σχέδια προτάσεων. Θέλουμε αυτό το θέμα να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Γερουσιαστά. Και τώρα, δώσ' το λόγο στην κυρία Πάιν. Φαντάζομαι θα σας διασκεδάσει τις εμφιβολίες και τους φόβους όσον αφορά τα σχέδια κανονισμού τα οποία θα περάσουν ή πέρασαν σήμερα στην ομική Επιτροπή όσον αφορά τα περιουσιακά των ε, συζύγων. Βεβαίω και η συζήτηση ήταν μακρά και έπρεπε κανείς να παρισχύσει για να πείσει τους ε, εμπλεκομένους. Όσον αφορά τα εθνικά συστήματα, τα οποία όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά ενισχύονται. Να πω και κάτι άλλο σε σχέση με όσα ακούσαμε από τον γερουσιαστή της, ε, της Πολωνίας. Είναι δεικτικό αυτό για το πόσο χρειάζεται κοινωνική ρύθμιση. Δυστυχώς που όμως δεν υπάρχει αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα οικογενειακού δικαίου. Το Κοινοβούλιο θα ήθελε πάρα πολύ να υπάρξουν ρυθμίσεις όσον αφορά τους ε, συζύγους, όσον αφορά την επιμέλεια των παιδιών, ε, γενικά τις γαμικές διαφορές και το διαζύγιο. Και να μπορούσε επομένω να υπάρξει εναρμόνιση των ρυθμίσεων που να ισχύουν επομένω κάποια πράγματα σε όλε τι χώρε. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στην Αλεξάνδρα, ε, μήπω κάποιο άλλο θα θέλει το λόγο ή να έχει να βρει κάποιε ερωτήσει. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένω, η σκητάλη στην Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ τους δύο συναδέλφους για αυτά τα οποία είπαν. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Ο κύριος Λέχνερ το είπε και στην αρχή. Όσο πιο πολύ ασχολείται κανείς με την ένωμη τάξη των διαφόρων κρατών μελών, διαπιστώνει πόσο διαφορετική είναι η μία από την άλλη, ειδικά σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου. Γι' αυτό θεωρώ, όπως και ο κύριος Λέχνερ, πως δεν μπορούμε να το εναρμονίσουμε όχι τις επόμενες δεκαετίες τουλάχιστον. Τι ήμουν πιο αισιόδοξη πριν έρθω εδώ πέρα. Και εγώ είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα και συμβολεογράφος, οπότε υπογράφω και έχω συντάξει πολλές ε, συμβάσεις ε, σχετικές ε, και συμβολεογραφικές πράξεις διασυγείου κτλ. Και νομίζω και ο κύριος Λέχνερ θα πει κάτι ξανά για το κληρονομικό δίκαιο. Οπότε κατά κανόνα δεν επεμβαίνουμε στο εθνικό δίκαιο. Μιλάμε εδώ πέρα για, τις, για τη ρύθμιση εκείνων των περιπτώσεων όπου δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε ευθύ αμέσω όταν ε, χωρίζει ένα ζευγάρι, ποιο, δεν μπορούμε να αμέσω ποιο δικαστήριο έχει αρμοδιότητα. Γιατί μπορεί κάλλιστα να ζουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, π.χ. ζούσαν μέχρι τώρα στην Ιταλία, χωρίζουν και ο ένας φεύγει και πάει, ξέρω εγώ, στην Πολωνία. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα ο ένας να πάει στα δικαστήρια στην Ιταλία και ο άλλος στην Πολωνία. Και Τώρα δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρεια το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Γιατί βεβαίως συμβολογράφη ολούμε κατά κύριο λόγο με τα κίνητα, αλλά θεωρητικά εάν πήγαιναν και οι δύο σε ένα δικαστήριο στη χώρα ε, προέλευσής τους θα μπορούσαν να εκδοθούν δύο διαφορετικές αποφάσεις με διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή το Ιταλικό Δικαστήριο να πει πώς ε, εφαρμόζεται εδώ πέρα το Ιταλικό Δίκαιο και το Πολωνικό Δικαστήριο να πει εφαρμόζεται εδώ το Πολωνικό Δίκαιο. Και δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό, έχει προσφύγει κανείς στα δικαστήρια, έχει εξοδέψει λεφτά, βγαίνει με απόφαση από την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα. Οπότε, αυτό που προσπαθούμε να λύσουμε. Τέτοιες περιπτώσεις ο καθένας, δηλαδή κάθε ζευγάρι, να γνωρίζει ε, εκ των προτέρων ε, και επίσης ε, ε καταχωρημένοι σύντροφοι στην περίπτωση στην οποία αυτό υπάρχει, να γνωρίζει εκ των προτέρων τι ισχύει, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στην περίπτωσή τους, να δοθεί δηλαδή στο κάθε ζευγάρι δυνατότητα επίσης ή δυνατότητα να επιλέξει εντός ορίων πάντα, έτσι. Αυτό ήταν, αυτό είναι τελικά το αντικείμενο εδώ πέρα. Και ε, στην περίπτωση τώρα που μιλάμε για κράτη που δεν έχουν τον θεσμό του συμφώνου συμβίωση ή κάτι, κάποιο ανάλογο δεν τίθεται ζήτημα α, αναγνώρισης του θεσμού, αλλά αν, ναι, μόνο των αποφάσεων άλλης χώρας. Π.χ. αν ένα ζευγάρι από το Βερολίνο πάει παραδείγματος χάρη στην ε, Πολωνία να εργαστεί. Οι πολωνικές αρχές, οι ε, δικαστήρια απλά θα αναγνωρίσουν πως το ζευγάρι αυτό έχει μια καταχωρημένη σχέση στη Γερμανία. Τίποτα περισσότερο. Γιατί ε, αυτή την στιγμή τι θα συμβεί τους λένε πως δεν έχουμε εμείς αυτό τον θεσμό του γάμου του ιδίου φίλου και υπάρχει νομίζω μια απόφαση και στο 10 ένα ισπανικό ζευγάρι πάει σε ένα άλλο κράτος μέλος και τους λέει μπορεί να είστε εσείς παντρεμένοι στην Ισπανία, ε, δύο γυναίκες ήταν, αλλά για εμάς ε, απλά μένετε μαζί. Και αυτό οδηγεί σε πρακτικά προβλήματα, έτσι, όταν ε, υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά δεν μπορούν να γραφτούν στον υπηαγωγείο, στο σχολείο, γιατί ο ένας από τους δύο γονείς δεν αναγνωρίζεται ως γονιός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν ξεκρέμαστα τα παιδιά. Εκεί όπου υπάρχουν παιδιά λοιπόν χρειάζονται πρακτικές λύσεις. Δεν, δεν γίνεται αλλιώς. Και δεν είναι δυνατόν μια άλλη περίπτωση πραγματική σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ε, στην Πορτογαλία νομίζω γεννήθηκε ένα παιδί και η Πορτογαλία λέει με συγχωρείτε κοιτάξτε τώρα είναι τόσο πολύπλοκες οι σχέσεις αυτές γιατί δεν ξέρω με ποια μέθοδο τεχνητής ε, γονιμοποίησης ή υιοθεσίας προήλθε το παιδί και δεν μπορώ εγώ να ξέρω τι υπηκότητα έχει το παιδί και πρέπει να μου το αποδείξετε εσείς και μετά σε δύο-τρία χρόνια θα κρίνω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και θα περιμένει δύο-τρία χρόνια το παιδί να αποκτήσει διαβατήριο. Και δεν μπορούν να πάνε οι γονείς ε, να ταξιδέψουν. Ε, γνωρίζουμε λοιπόν πως είναι τελείως ε, πρακτικά τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν τα χαρτιά τους ε, δύο-τρία χρόνια και να ταξιδεύουν με το παιδί, να μην φαίνεται ότι το παιδί είναι δικό τους. Δεν αναγκάζουμε λοιπόν πολωνικό ή ιταλικό δικαστήριο να πει, να αναγνωρίσει σχέσεις, ε, μάλλον γάμους ή σύμφωνα του ιδίου φίλου. Απλά να γνωρίζετε πως ε, υπάρχει αυτή η σχέση σε μια ε, άλλη χώρα. Και από τα ζευγάρια αυτά λέμε πως δεν έχει προχωρήσει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάτε είτε στο, στη χώρα, σε ένα δικαστήριο στη χώρα όπου έχετε επισημοποιήσει τη σχέση ή κάπου όπου ισχύει έχουν στην ένωμη τάξη τους ε, τον γάμο των ομοφιλοφίλων για να λυθεί εκεί ο γάμος. Γι' αυτό ε, γιατί βεβαίω θα μπορούσε κανεί να σκεφτεί, άμα τα αναγνωρίζετε στου ξένου, θα τα αναγνωρίζετε και σε εμά. Πώ αλλιώ. Ε, για να αποφύγουμε λοιπόν ε, αυτό, έχουμε βάλει τόσε πολλέ περικοκλάδε και δικλείδε ασφαλεία στο κείμενο για να ξεκαθαρίσουμε πω δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλά ισχύει μόνο σε περιπτώσει με διασυνοριακό χαρακτήρα και ε, όταν αφορά όπως είπα, τέτοιες ε, περιπτώσεις. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα απέτησης ε, Πολωνού πολίτη έναντι του πολωνικού κράτους. Να καταχωρηθεί μια τέτοια σχέση, ας πούμε. Και... Όσον αφορά τώρα τα παιδιά και ποιος θα πάρει τα παιδιά, αυτό δεν το ρυθμίσαμε καθόλου. Και γιατί μετά θα μπούμε και σε ζητήματα διεθνούς απαγωγής ε, και τα λοιπά. Οπότε ισχύουν μετά άλλες καταστάσεις. Π.χ. στο γερμανικό δίκαιο πάνε τα παιδιά στο, στο γερμανό γονέα. Και δεν, κοιτάξτε, δεν ε, έχω λοιπόν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία σε περιπτώσεις που έχουμε ένα γάμο με δύο εθνικότητες και σε ποιον πάει στον άλλο. Αυτό μου το είχαν καταγγείλει, δεν ξέρω αν ισχύει όντως ε, και αν ε, εφαρμόζεται αυτό κατά κανόνα. Οπότε από συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως φαίνεται να δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Αλλά ισχύει και το αντίθετο. Υπάρχουν δηλαδή και Γερμανοί οι οποίοι παραπονούνται πως δώσανε σε άλλο κράτος στον γονέα του οικίου με την οικία επικοότητα το παιδί. Και το ίδιο παράπονο κάνουν οι Γάλλοι για εμάς τους Γερμανούς. Ε, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ισχύει όντω για να το κάνουν αυτό τα δικαστήρια. Θα πρέπει κάποια στιγμή πάντως να δούμε τα στατιστικά στοιχεία, να δούμε αν ισχύει πράγματι αυτό το οποίο λένε οι πολίτες, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις. Τώρα σε τρίτες χώρες να πάρουν τα παιδιά και να τα δώσουν σε ανάδοχη οικογένεια, αυτό δεν το είχα ξανακούσει. Αλλά... Το πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και μας απασχολεί στην ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δηλώσει για κάποια κράτη-μέλη πως ε, ε, έχουν προσχωρήσει στην ε, συνθήκη της Χάγης ή αν ε, πρέπει να το κάνει το ίδιο το κράτος, αν δηλαδή θα πάει μέσω κοινοβουλίου ή συμβουλίου. Αλλιώς με όλο αυτόν τον τομέα δεν έχουμε ασχοληθεί. Όσον αφορά δε τον, το θέμα της διατροφής, εάν ο πατέρας κατά κανόνα, αλλά καμιά φορά και η μητέρα οφείλει να πληρώσει διατροφή και δεν πληρώνει. Αυτό το ρυθμίσαμε μέσω της κεντρικής υπηρεσίας σε κάθε κράτος που θα βοηθά τον κάθε γονέα για τις απαιτήσει του έναντι του άλλου. Αλλά τίποτα περισσότερο, τίποτα περισσότερο δεν ρυθμίσαμε, καμία άλλη αρμοδιότητα δεν δώσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Η Αλεξάνδρα απάντησε στα σχόλια των εκπροσώπων των κρατών μελών. Και από την απάντησή της φαίνεται πόσα εργοτάξια αστικού οικογενειακού δικαίου ε, έχει να ολοκληρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα θα δώσουμε τα, το λόγο στον κύριο Λέχνερ για να πει δύο λόγια για τις κληρονομιές. Και μετά σιγά σιγά θα κλείσουμε. Ναι. Ο Ιταλός συνάλφος πρέπει να προλάβει το αεροπλάνο και έφυγε. Να πω λίγα ποια πράγματα για την αμοιβή αναγνώριση και για τους νομικούς εδώ εντός εύσως το γλωσσικό ζήτημα και η μετάφραση ήταν ουσιαστικό γιατί βεβαίως πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβείς οι εκφράσεις και είχαμε συνεχώς προβλήματα με την ε, μετάφραση και βεβαίως ε, το θέμα της ε, αμοιβαίας αναγνώρισης δεν είναι προβληματικό πολιτικά αλλά κοιτάξτε παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών, η πρόταση Κομισιόν ήταν ε, τελείως ε, χοντροειδής. Κάνουμε μια μετάφραση και τελείωσε. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένα τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση αυτό, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Αλλά αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ τότε στην Επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος Μπερλίνγκουερ ε, ως εισηγητής των σοσιαλιστών ε, από την Ιταλία. Το ότι δηλαδή εμείς δεν θέλαμε υπό, σε καμία περίπτωση να περάσουμε στο ουσιαστικό κληρονομικό δίκαιο των κρατών μελών. Βεβαίως αυτό εύκολα το λέει κανείς αλλά δύσκολα γίνεται. Γιατί ε, διαφέρει και το εύρος και το πεδίο εφαρμογής των, του κληρονομικού δικαίου. Και εντάξει, αυτά ήταν, δηλαδή που σταματάει το δικονομικό και που αρχίζει και το ουσιαστικό δίκαιο στην περίπτωση αυτή. Αλλά όπως είπα στα κράτη-μέλη έχουμε Έχουμε δύο τελείως ρυθμίσει ε, ρυθμίσεις ε, όσον αφορά την Ιταλία, Αυστρία, Ιταλία, π.χ. το τι γίνεται με την ε, νόμιμη μοίρα των συζύγων και των λοιπόν και αν υπάρχει καν νόμιμη μοίρα σε πολλές περιπτώσεις. Ε, και διαφορετική κατάσταση στη Γερμανία και όλα αυτά έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Το να γίνει αυτό θα οδηγούσε αφενός σε ζητήματα νομικής ασφάλειας και όταν έκανε κάποιος το, τον προγραμματισμό του, όταν συνέτασε την ε, διαθήκη του και θα πηγαίναμε σε μια λύση που θα ήταν ανάλογη με αυτή που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, όπου το Ιταλικό δίκαιο αναγνωρίζει. Υπάρχουν π.χ. πάρα πολύ κάτοχοι εστιατορίων, πιτσεριών που για να αφήσουν το εστιατόριο επιλέγουν το γερμανικό δίκαιο. Κατοικούν στην Γερμανία και ε, μετά λένε υπό την επιφύλαξη των όσων λέει το Ιταλικό Δίκαιο για την ε, νόμιμη μοίρα. Οπότε, τι γίνεται σε αυτή την ε, περίπτωση. Η αναγνώριση λοιπόν του τι προβλέπει το κληρονομικό δίκαιο μιας άλλης ε, χώρας, ε, του Ιταλικού ή του Γαλλικού, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί, δημιουργεί ένα πρόβλημα γιατί είναι κάπως πιο ελαστικό, εάν θέλετε, το γερμανικό δίκαιο σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Να μιλήσω για την ε, Μεγάλη Βρετανία, όπου δεν τίθεται ζήτημα νόμιμης μοίρας σε ε, Αγγλία και Ουαλία. Και <coughs> αν κάποιος μεταφέρει όλη του την περιουσία, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, δεν δεν υπάρχει καν ε, τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, και μπορεί βεβαίω να πάρει μια απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση, ένα Ιταλικό δικαστήριο, η οποία όμω δεν αναγνωρίζεται μετά στην Αγγλία, έτσι. Δεν αρκεί να μεταφέρει επίσης κάποιος ε, τα περιουσιακά του στοιχεία ή και την κατοικία του σε μια χώρα, πρέπει να παραμείνει εκεί και επίσης να αποβιώσει εκεί πέρα. και ε, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο βέβαια απέτυχε και οποιοδήποτε συνδυασμός με την ε, Μεγάλη Βρετανία. Και να σας πω πως, ε, κοιτάξτε και εγώ προσωπικά δεν είμαι παδός τόσο μεγάλος της νόμιμης βίρας, αλλά δεν είναι και η αρμοδιότητά μου, έτσι, ούτε είναι δουλειά μου να μπαίνω εγώ στα χωράφια αυτά. Αλλά στην ε, Μεγάλη Βρετανία υπήρχε το λεγόμενο clawback. Ε, το πότε το... Το, βρήκα. το, ζήτημα είναι λοιπόν πως ε, τώρα ήταν διάφορα ζητήματα με το να μην μπορεί κανείς να διεκδικήσει να μπορεί κανείς να κάνει τίποτα στην περίπτωση που είχε εγκατασταθεί ο παθανόν στην ε, Αγγλία. Οπότε, τι έχουμε στην περίπτωση που ένας Ιταλός, Γερμανός ε, ή Άγγλος ε, πήγαινε στην Αγγλία και μεταφέρει εκεί πέρα την περιουσία του. Ε, για αυτό το κομμάτι, αν έμπαινε μέσα η Αγγλία, για αυτό το κομμάτι της περιουσίας του που είχε μεταφέρει θα ίσχυε στην ε, Αγγλία ένα δικαίωμα το οποίο δεν ε, αναγνωρίζουν κανονικά. Και μην ξεχνάμε τι γίνεται και στην ε, περίπτωση στην οποία κάποιος ε, γιατί στην οποία κάποιο Γάλλο, α πούμε από το Στρασβούργο πάει και μετακομίζει στο ΚΕΛ. Έχουμε και το θέμα τη ε, προθεσμία των 10 ετών η οποία ισχύει συχνά. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κοντά η Γερμανία με την ε, Αγγλία σε αντίθεση με την Γαλλία η οποία η Γαλλία και η Ιταλία έχουν πάρα πολύ αυστηρό ε, δίκαιο στο ζήτημα της νόμιμης μοίρας, ενώ μετά από κάποια χρόνια δεν τίθεται ζήτημα τέτοιο στην ε, Γερμανία και όπως είπα καθόλου στην Αγγλία. Επειδή λοιπόν θα μπαίναμε πάρα πολύ στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, ε, είπαμε πως ε, δεν θα μπούμε σε αυτό το ζήτημα. Γιατί εντάξει δεν υπάρχει μόνο η Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν τρίτες χώρες, μουσουλμανικές χώρες όπως το Μαρόκο που επίσης είναι αντικείμενο. όπου εκεί πέρα κληρονομούν οι, γη και κληρονομούν τα διπλά από τις κόρες. Έτσι αυτό κατά την άποψή μου παραβιάζει νομίζω το, το δικό μας το, το δίκαιο. Και Υπάρχει νομίζω και μία απόφαση σχετική ενός ε, γερμανικού δικαστηρίου που είχε πει πως ε, ε, αν ήθελε ο, Μαροκανός, ο Μαροκινός πατέρας θα μπορούσε να κάνει τον γιο του μοναδικό κληρονόμο και θα έλαμβανε την νόμιμη μοίρα η κόρη μετά που της αναλογούσε και μάλιστα σε λεφτά όχι σε είδος. Αλλά εφόσον δεν έκανε τίποτα θα τα μοιραστούν στα δύο και ε, τελείωσε. Με το να μην κάνει δηλαδή τίποτα ο πατέρας τελικά πήρε κόρη περισσότερα από όσα θα της έδινε σε αντίθετη περίπτωση οπότε τελικά δεν παραβιάστηκε το δίκαιο του... της Γερμανίας συγκεκριμένη περίπτωση. αλλά όπως σας είπα δεν ε, μπήκαμε σε αυτό το ζήτημα γιατί θα, όπως βλέπετε τα ζητήματα που ανακύπτουν είναι πάρα πολλά και θα ανοίγαμε πάρα πολλά μετά. Ευρωπαίοι πολίτες ε, οι οποίοι πάνε σε μια άλλη χώρα, ζουν, ε, εργάζονται και πεθαίνουν, εντάξει, λογικό είναι να ισχύσει το τοπικό δίκαιο κάθε φορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λέχναρ την κυρία Φιωρίνη. Την ευχαριστήσουμε, αλλά επίσης και την κυρία Τάινη. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο ε, από την Νομική Επιτροπή, τον κύριο Λουίτζι Μπερλιγκουέρ. Και τώρα, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας συζήτησης και θα συζητήσουμε τα εργαλεία που έχουμε για μια, αποτελεσματική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου τον κύριο Λέχνερ, που τον ακούσατε να μιλάει λίγο πριν από μένα. Εξαφανίστηκε τώρα, έφυγε. Δεν πειράζει όμως. Ο Λέχνερ ήταν ευρωβουλευτής μέχρι πριν από ένα χρόνο και ήταν εισηγητής για θέματα κληρονομιάς. Ήταν μια απίστευτη ιστορία αυτή, χρονοβόρα, δύσκολη, κουραστική, όπως πάντα είναι τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα, αλλά αυτό ήταν εξόχως κουραστικό και χρονοβόρο. Γιατί άγγιζε την καρδιά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και έπρεπε να συγκεράσουμε διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές πραγματικότητες, αν θέλετε, των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Γιατί δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο όλοι πεθαίνουν κάποια στιγμή και πολλοί, αν όχι όλοι, αφήνουν μια κληρονομιά πίσω τους. Επομένως, αυτό ήταν ένα από τα νομοθετήματα που άγγιζε την καρδιά της Ευρώπης. Ναι, και οι παραδόσεις γι' αυτό είναι πολύ διαφορετικές. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο συνάδελφος αυτός, ο φίλος, ο κύριος Λέχνερ, δούλεψε με τέτοιο πάθος, με τέτοια υπομονή και υπομονή για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, γιατί τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα είναι πάντα καρπός υπομονής, υπομονετικής δουλειάς μέχρι το τέλος. Αυτή η δουλειά χρειάστηκε να γίνει λόγω των διαφορών που έχουμε στα διαφορετικά κράτη-μέλη, λόγω των φοβερών αντιστάσεων που έχουμε, της προσκόλλησης της παραδόσης μας και του γεγονότος ότι, και αυτό το λέω στρέφομαι κυρίως προς εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, Θέλω να σας πω ότι εμείς οι νομοθέτες, ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές, έχουμε ένα μεγάλο πάθος και αρεσκόμαστε στον νομοθετήν. Αλλά δεν έχουμε το ίδιο πάθος στο να παρακολουθούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ενεργοποιηθεί η νομοθεσία. Πώς εφαρμόζεται δηλαδή και πώς ζουν τα αποτελέσματα αυτής της νομοθεσίας οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τι εντύπωση έχουν, τι συμβαίνει. Γιατί πολύ συχνά συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε γράφοντας ένα νομοθέτημα. Γιατί στην πραγματικότητα απλώς εμείς αντιδρούμε. Και πρέπει λοιπόν στην νομοθετική δουλειά να μάθουμε, να διδαχτούμε. Δεν είναι μόνο, το θέμα δεν είναι μόνο να παράγουμε νόμους, αλλά να είναι λειτουργική αυτή η νόμη. Και θα πρέπει ε, η τροχιά αυτών των νόμων να έχει επαφή με την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν στατιστικές που λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα νομοθετικό κόρπους, ένα κόρπους γιούρις, απίστευτο, εντυπωσιακό, τιτάνιο, αλλά μόνο το 5% των πολιτών, σε, τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς, εποφελείται από αυτό το κόρπους. Είναι σαν να αγοράζει Φεράρι και να τρέχεις με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν δικαιολογείται η προσπάθεια. Αν εμείς δεν δουλεύουμε και για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ούτω ώστε αυτό που φτιάξαμε στην νομοθεσία να απορροφάται από την κοινωνία και να βιώνεται από την κοινωνία, δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί είναι και αυτό το τμήμα της νομοθεσίας. Σήμερα λοιπόν εμείς σε αυτό το τέταρτο πάνε θα πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας. Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν κοινή δικαστική κουλτούρα όλοι οι Ευρωπαίοι δικαστέ έχουν μία ιδέα για τη δικαιοσύνη και αυτή η ιδέα είναι ίδια. Μία ε, διοντολογία που είναι ίδια. Μία ιδέα για την ε, λειτουργία των, α, ε, της δικαιοσύνης που είναι ίδια. Απλώς είναι διαφορετικές οι δικαστικές παραδόσεις. Εμείς ζούμε στη μοναδική ένωση και εμπειρία μας από την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δείχνει ότι η Ευρώπη γίνεται ένα χωνευτήρι, όπου οι διαφορετικές παραδόσεις και πάνω απ' όλα ε, η παράδοση του, των χωρών του common law, παρότι διατρέχει τελείως διαφορετικό δρόμο, ακόμα και τα ονόματα αρχίζουν να αλλάζουν και να συγκλίνουν με τις υπόλοιπες Ευρώπης. Θυμάμαι πόσο δύσκολο ήταν να μεταφράσουμε στα αγγλικά το νομική προσωπικότητα. Εγώ είμαι Ρωμαίος, πολίτης, ξέρω το ρωμαϊκό δίκαιο και δεν ήξερα πώς να το μεταφράσω αυτό στα αγγλικά. Σήμερα ακούμε τον όρο legal personality. Στην αρχή, παλιά ήταν αυτό λάθος, αλλά τώρα μπαίνει στην αγγλική γλώσσα. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι δημιουργική και στο επίπεδο της κουλτούρας αυτή η, η γάμη, αυτή η πολυγαμία, των 20, δηλαδή το πάντρεμα των 27 διαφορετικών ένομων τάξεων δίνει αποτελέσματα. Επομένως, από τη μία, έχουμε την κατάρτιση των δικηγόρων, να μην το πω εκπαίδευση, γιατί είναι ήδη εκπαιδευμένοι αυτοί οι άνθρωποι, που η κατάρτιση στην πραγματικότητα είναι εξέλιξη περισσότερο. Η κατάρτιση λοιπόν των δικαστών, Φερρυπίν, πρέπει να μας απασχολήσει και να δούμε τι μορφή πρέπει να πάρει αυτή η δραστηριότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον δύο φορές αποφάνθηκε με επίσημα έγγραφα στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης και μιας άλλης πρωτοβουλίας, με πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για αυτό το θέμα, με σκοπό να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα. Αυτός είναι πάντα ο στόχος. Ε, υπενθυμίζουμε μια μεγάλη α, Ολλανδέζικη εμπειρία σε αυτά τα κείμενά μας. Ο, ο Ρουντ είναι ένας από τους δημιουργούς αυτής της Ολλανδικής εμπειρίας. Επίσης, θα πρέπει να συγκρίνουμε διάφορα συστήματά μας, ούτω ώστε να κρατήσουμε υψηλό επίπεδο. Μην ξεχνάμε τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, όπου οι εθνικοί δικαστές είναι ταυτόχρονα και Ευρωπαίοι δικαστές. Με αυτό το Justice Scoreboard, ο πίνακα αποτελεσμάτων για τη δικαιοσύνη, μπορεί να βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κλείνοντα, θέλω να πω ότι αν θέλω να προωθήσουμε όχι μόνο το νομοθετήν, αλλά και την εφαρμογή τη νομοθεσία, ένα από τα εργαλεία για να το επιτύχουμε είναι το εργαλείο της κοινή ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας. Μετά τα αυτά θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ρουτ Βίντερ, ανώτατος αντιπρόεδρος συντονιστής του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου για εμπορικές και βιομηχανικέ υποθέσεις, υποθέσεις των κάτω χωρών. Στην Ολλανδία. Είναι τιμή και προνόμιο το να βρίσκομαι εδώ, στην καρδιά της Ευρώπης, για να σας, μιλήσω, ε, να σας πω διάφορα πράγματα για τη δημιουργία δικτύων για την κατάρτιση σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Θα σας δώσω πολύ σύντομα ε, κάποια στοιχεία για την επαγγελματική μου το επαγγελματικό μου παρελθόν. Επί 25 χρόνια δούλεψα ως εθνικός ε, Ολλανδός δικαστής που ασχολήθηκα με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου ένας δικαστής στην Ολλανδία πρέπει να ασχολείται συνέχεια με το ευρωπαϊκό δίκαιο όταν ασχολείται με γεωργικά θέματα, θέματα τροφίμων, ε, λιπάσματα, ζανιοκτώνα κτλ. Ήμουν δηλαδή δικαστής, πραγματικά ευρωπαϊκός δικαστής, ε, στον προμαχώνα της Ευρώπης. Η θέση μου στο δικαστήριο μου επέτρεψε όχι μόνο να αποκτήσω μια μεγάλη εμπειρία εφαρμόζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά πολλές φορές είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε προγράμματα στα πλαίσια της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για να μοιραστώ την εμπειρία μου με άλλους ομολόγους δικαστές διαφορετικών κρατών μελών. Σε αυτές τις συναντήσεις είχα την ευκαιρία να ακούσω τις επιθυμίες τους, τις ανησυχίες τους για το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις παρατηρήσεις τους που τη συνοψίζω ω εξή. Πού να το βρω αυτό, πώς να το χρησιμοποιήσω, υπάρχει εργαλειοθήκη, υπάρχει οδηγό που μπορεί να με βοηθήσει. Στην Ολλανδία η εμπειρία μου με το θέμα αυτό ξεκινάει από το 2001, όπου είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω να συμμετάσχω σε ένα πρόγραμμα όπου Ολλανδοί δικαστές συμμετείχαν γιατί θεώρησαν ότι δεν είχαν αρκετή γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Υπουργό ε, Δικαιοσύνη ε, διέταξε να αλλάξει αυτή η κατάσταση, η άγνοια δηλαδή, του ευρωπαϊκού δικαίου, το συντομότερο δυνατόν. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε γνώση ε, για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μιλάμε ε, για την κατάρτιση δηλαδή μη ειδικών δικαστών που έπρεπε να βρουν και να εφαρμόσουν κάθε τόσο ας πούμε μια στο τόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή ο μέσος δικαστής. Και βασιστήκαμε σε τρεις πυλώνες. Να βελτιώσουμε την προσπελασιμότητα του ευρωπαϊκού δικαίου χρησιμοποιώντας την πληροφορική, δηλαδή δημιουργήσαμε το, τη δικτυακή πύλη Euris και τη δικτυακή πύλη Ευρωπαίου, ούτως ώστε να μάθουν καλύτερα το ευρωπαϊκό δίκαιο οι Ολλανδοί δικαστές, χάρη στη μεγαλύτερη κατάρτιση, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο όπου δικαστές όλων των δικαστηρίων της Ολλανδίας γράφαν σε ένα blog. Και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Το γενικό συμπέρασμα από την εμπειρία μας ήταν ότι αυτή η δομή σε τρεις πυλώνες ήταν πολύ αποτελεσματική και άντεξε στο πες του χρόνου. Ακόμα και σήμερα είναι επίκαιρο το ερώτημα του πού θα βρω την σχετική χρήσιμη πληροφορία. Δεύτερος πυλώνας. Ε, γνώσεις και δεξιότητες για να χρησιμοποιήσω την γνώση. Πότε να εφαρμόσω το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κατάρτιση είναι η λέξη κλειδί εδώ. Ο τρίτος πυλώνας ε, δημιούργησε μια λυσίδα από αφοσιωμένους επαγγελματίες που χρησιμεύαν ως ε, blogger που ήξεραν τα πράγματα και αποτελούσαν το σημείο επαφής μεταξύ των δικαστών. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ευέλικτο δίκτυο που μας ε, επέτρεψε να ε, δεχόμαστε ερωτήσεις και να δίνουμε γρήγορες απαντήσεις. Αυτό που ήταν πάντα και είναι σημαντικό είναι ότι η δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας σε ένα πυλώνα πάντα πρέπει να εντάσσεται ε, στο εσωτερικό της δομής αυτού του προγράμματος, του δικτύου και να συντονίζεται με τις δραστηριότητε των άλλων πυλών. Έτσι λοιπόν ο Ολλανδός δικαστής, υπάρχει ένας Ολλανδός δικαστής που έχει συντονιστικό ρόλο. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι δικαστές και οι επαγγελματίες της δικαιοσύνης λειτουργούν σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό. Όταν κοιτάμε την πραγματικότητα σήμερα, βλέπουμε ότι την τελευταία δεκαετία η τεχνολογία έκανε ένα απίστευτο βήμα προ τα εμπρό. Η πρόσβαση των πληροφοριών, πληροφορίε, ε, είναι πολύ πιο εύκολη σε όλου του τομεί τη ζωή. Η προσπέλαση της, του ευρωπαϊκού δικαίου είναι πολύ πιο εύκολη επίση και για του Ολλανδούς δικαστέ. Η βελτίωση τη ε, τεχνολογία στον πρώτο πυλώνα εξασφάλισε την προσπέλαση τη πληροφορία και μα αναγκάζει να επανεξετάζουμε τη σχέση που έχει ο πρώτος πυλώνας με το δεύτερο πυλώνα, προκειμένου να λειτουργήσει καλά το δίκτυο συντονιστών του τρίτου πυλώνα. Ε, η αρχική δομή, η αρχική αρχιτεκτονική του προγράμματος η, ακόμα είναι σε λειτουργία. Απλώ το περιεχόμενο αλλάζει, δηλαδή η αρχιτεκτονική παραμένει, το περιεχόμενο αλλάζει. Επαναλαμβάνω, η κατάρτιση είναι πολύ βασική. Ε, Πληροφορίε πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμες και τότε όταν συμβαίνει όμω αυτό η κατάρτιση μπορεί να ε, διαρθωθεί με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Η, η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε με πολύ περισσότερους τρόπους. Ε, e-learning με online μαθήματα, είναι απλώς λίγα παραδείγματα. Τα δίκτυα είναι πάντα πολύ σημαντικά και μπορούν να λειτουργήσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι παλιότερα. Επομένως, ξεφύγαμε από το παρελθόν και μπαίνουμε σε ένα τελείως νέο περιβάλλον τώρα, σε μια νέα εποχή. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι όταν πρέπει να θες να συνθέσεις μια ωραία μελωδία, πρέπει να έχεις όλες τις νότες στη διάθεσή, του, στη διάθεσή σου και στη σωστή θέση. Για να μπορέσουν οι μουσικοί να δώσουν στον κόσμο να καταλάβει και να νιώσει την ουσία της μουσικής. Αυτή είναι η ουσία της μουσικής. Στην ε, τεχνολογία ε, τα δίκτυα θα πρέπει να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε η κατάρτιση να εξασφαλιστεί αμέσως βάση και χάρη στην εύκολη πρόσβαση της πληροφορία που παρουσιάζεται με πολύ εύληπτο και λογικό τρόπο. Τα δίκτυα λοιπόν εποφελούνται από τα ωφέλη των μοντέρνων τηλεπικοινωνιών και να ε, εξυπηρετήσουν τους στόχους, να δώσουν πληροφορίες, να ενημερώσουν για τις νέες εξελίξεις σε πρώιμο στάδιο ήδη. Ο συνδυασμός λοιπόν της έλλειψης χρόνου που συχνά ακούμε από τον κόσμο σήμερα, έλλειψης χρημάτων, ακόμα πιο πολύ το ακούμε αυτό, και της πολύ καλής τεχνολογίας, ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να θεωρηθεί η καρδιά και η ατμομηχανή της ε, προσπάθειας για εξασφάλιση της πρόοδου μέσα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Σήμερα συχνά βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου η πληροφορία, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και τα δίκτυα δεν θεωρούνται διαφορετικοί πυλώνες του ίδιου κτηρίου. Οι σημειώσεις δηλαδή δεν είναι πάντα σωστά παρμένες. Ε, οι νότες, οι μουσικές νότες δεν βρίσκονται σωστά στο πεντάγραμμο, επομένως δεν μπορούν να καταλάβουν οι μουσικοί πώς μπορούν να αποδώσουν ωραία τη μουσική. Και έτσι λοιπόν συχνά το ακροατήριο φεύγει από την αίθουσα... Πες το Τη συναυλίας πολύ δυσαρεστημένος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της κατάρτισης των ε, Ευρωπαίων δικαστών. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο τρόπο την ύπαρξη των διαφόρων δικτύων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου. Το σκεφτόμουν λοιπόν αυτό και προσπαθώ να σκεφτώ πώς, ε, τι μορφή θα έχει το επόμενο δίκτυο. Το δίκτυο στο μέλλον δηλαδή. Θα πρέπει να έχουμε πληροφορία, κατάρτιση, δίκτυα. Θα πρέπει επομένω αυτά να αναγνωρίζονται ω οι πυλώνε του συστήματο και με συνεργασία και συντονισμό ε, μεταξύ αυτών των πυλώνων είναι πάρα πολύ αναγκαίο και κάθε ε, ε, νομικό θα μπορεί να βρει την πληροφορία που του χρειάζεται. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστε αυτέ οι πληροφορίε και θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένοι και θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα εύκολη και να είναι εύκολο το σύστημα. Αυτό επομένω η πύλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι η πύλη σε όλε τι νομικέ πληροφορίε και να είναι όλα επιχειροποιημένα. Η εκπαίδευση χρειάζεται για να υπάρχει ευρύτερη γνώση και καλύτερη και ποιοτικότερη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε την ε, ανταλλαγή εμπειρίας. Όταν είναι εύκολα προσβάσιμες οι πληροφορίες, τότε θα πρέπει αυτή η κατάρτιση να προσαρμόζεται σε αυτή την νέα κατάσταση. Διαφορετικές μορφές, διαφορετικά εργαλεία ε, και λιγότερο χρονοβόρια διαδικασία. Θα πρέπει να γίνεται τέτοια κατάρτιση face to face, οπότε να μπορούμε να ευνοήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Αυτό το δίκτυο θα πρέπει ακριβώς να κατατείνει ε, σε τέτοια εκμετάλλευση αυτής της πληροφορίας που να χρησιμοποιείται ε, από όλους και θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη από οποιοδήποτε σημείο. Να χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, του, ψηφιακού δικτύου, ούτως ώστε τα κράτη-μέλη με ασφάλεια να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι ρόδινο. Όλα αυτά πρόκειται να συνδυαστούν και να βοηθήσουν. Πολύ ελκυστικό θα είναι ε, αυτό το e-justice. Θα προσφέρει όλα αυτά που είπαμε, θα είναι φιλικό στο χρήστη και έτσι θα εξηγεί τα βασικότερες έννοιες του κοινωτικού δικαίου. Ιδιαίτερως αυτά χρειάζονται Κάθε φορά που αυτές οι αρχές πολλές φορές δεν ανεβρίσκονται στην ε, συνθήκη. Γιατί αυτές οι βασικές αρχές αναδύθηκαν από την νομολογία του 10. Οπότε θα περιγράφονται εκεί πέρα και κατανοητά για τους πολίτες και με λεπτομέρειε για τους νομικούς Και όλοι οι νομικοί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν πάρα πολύ εύκολα να έχουν πρόσβαση εκεί πέρα για ε, όλα τα θέματα του γενικού δικαίου. Πώς να το πείτε, εργαλείο και όπως ακριβώς έχουν ζητήσει οι συνάδελφοι δικαστές στα νέα κρατημέλη, αλλά δεν το ζητούν μόνο αυτοί αυτό το εργαλείο, την εργαλειοθήκη. Ίσως αυτό θα είναι μια θετική, μια επικοδομητική συμβολή ε, στην κατάρτιση των 700.000 νομικών. Όπω είπε, ανακοίνωση τη 13 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη το καθένα ε, θα πρέπει για κάθε νομικό να δώσουν 100 ευρώ. Άρα μιλούμε για 70 εκατομμύρια ευρώ που είναι ένα μικρό κλάσμα του το, ποσού που χρειάζεται για να έχουμε αυτή την ε, πλατφόρμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει μια γενική έποψη του τοπίου που ισχύει κάθε φορά για το κοινωτικό δίκαιο και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο διαδίκτυο προσφέρει πληροφορίε, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε το σύστημα α πούμε τη ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων, ένα σύστημα PowerPoint, μια παρουσίαση, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αξιολογήσουμε, να, για να εκμεταλλευτούμε αυτή την, ε, αυτή την πύλη. Και και μέσω του Google ε, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την πύλη. Δυστυχώς όμως όχι στην ομολογία του δικαστηρίου. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό με συνδέσμους. Όμως, αν κανείς πάει στο Google και ψάξει να βρει κάτι για την ελεύθερη ας πούμε διακίνηση εμπορευμάτων, δεν θα βρει αυτά τα οποία θα βρει στην, ε, στην πύλη τη διαδικτυακή αυτή της Κομισιόν. Τι θέλω να σας πω, ότι ε, τώρα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα μπρος όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ε, μπορεί κανείς να πάει εκεί πέρα στον σύνδεσμο που λέει νομολογία, θα βρει έναν ορισμό της λέξης νομολογία και η... Ε, όμως αυτό για τους νομικούς δεν ωφελεί πολύ αυτό και για τους υπολείπους. Τώρα πάμε κανείς στο Ρέλεξ, θα, θα βρει κανείς το αλφάβητο του κοινωτικού δικαίου. Όμως εκεί δεν υπάρχει η αναγκαία ακρίβεια και είναι και μπερδεμένα άλλωστε για τους πολίτες. Επομένως τελικά τα δίκτυα ε, βοηθάνε. Όπως προανέφερα. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι το πρώτο βήμα ούτως ώστε να προλυάνει κανείς το έδαφος για να έχουμε μια αποτελεσματική παιδεία. Οπότε πρόκειται επίσης για τις προϋποθέσεις ε, που συντρέχουν για αποτελεσματικό δίκτυο. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι ρόδινο για το κοινοτικό δίκαιο και γι' αυτό και θεωρώ ότι ανοίγει λεωφόρους πληροφοριών αυτή η πύλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ περισσότερα δίκτυα θα υπάρξουν από όσα υπάρχουν τώρα. Και τέτοιε εκπαιδευτικέ δραστηριότητε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο που μπορεί βεβαίω αυτό να θεωρείται ε, ένα μεγάλη πρόοδος γιατί μπορούμε έτσι ηλεκτρονικά να έχουμε ομιλίες, ε, συμπόσια και επίσης κάποια και μαθήματα που παρακολουθήσει κανείς να σπουδάσει οπότε έτσι βελτιώνει την κατάσταση για να έχουμε συντονισμό και να ξέρουμε τις δραστηριότητες που αποναντήσονται παντού. Τέτοια δίκτυα σε πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα όσο γίνεται περισσότερο. Ladies Κυρίες και κύριοι, για να προσγειωθούμε τώρα μετά από αυτές τις υψηλές σκέψεις θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι για την ε, κατάρτιση των δικαστών είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα δίκτυα άπαξ και μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Γι' αυτό και βλέπω ρόδινο το μέλλον για αυτά τα δίκτυα. Οπότε έτσι θα μπορούμε να δουλέψουμε ηλεκτρικά περισσότερο χωρίς αυτό να υποκαταστήσει την προσωπική επαφή. Όπως ακριβώς ε, και σήμερα που συνθήκαμε εδώ, γιατί όπως προείπα, το περιβάλλον στο οποίο οι νομικοί εργάζονται έχει αλλάξει πάρα πολύ και οι αλλαγές θα σταματήσουν σήμερα, θα σταματήσουν εδώ. Αλλά θα πρέπει και πάλι να σταθμίσουμε πληροφορίες, παιδεία και δίκτυα και επίσης ακριβώς όπως μια ε, ορχήστρα αποδίδει καλά ένα μουσικό κομμάτι, να μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα στους νομικούς να αποδώσουν όσο μπορούν καλύτερα. Να βγάλουν μια μελωδία που να αρέσει σε όλους και για το καλό όλων. Σας ευχαριστώ. Έφτασε και ο πρόεδρός μας, ο καθηγητής Ρόπερς Λόπες Αγγιλάρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βίντερ για τη θέση του και για την παρουσίαση που μας έκανε. Που υπογραμμίζει νομίζω ότι καμία διαδικασία κατάρτισης ή προώθησης της επαγγελματικής καριέρας του, των δικαστών των, ή των δικηγόρων δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς τη χρήση δικτύων και του ίντερνετ γενικά. Αν και τόνισε και τη σημασία των επαφών εκ του σύνεγγης, πρόσωπο με πρόσωπο. Χρειάζεται... Αλλά και οι διαδικασίες κατάρτισης και τα δίκτυα δεν μπορούν να θεωρηθούν εργαλεία ψυχρά και ουδέτερα. Προωθούν τις γνώσεις και την κατάρτιση και την πρόσβαση στη γνώση. Δεν είναι η γνώση αυτά καθεαυτά. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη γνώση που επιθυμούν. Η ομιλία του Ρουντ μου θύμισε αυτά που έλεγε ο Λούθυρος για τη δουλειά που γίνεται με καλό τρόπο. Έβαλε την ιδέα, εισήγαγε στο μυαλό μας την περηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν η δουλειά γίνεται καλά. Και ο Ρίτσαρτ Σένετ σήμερα μιλάει πάλι γι' αυτό στα βιβλία του. Και θα πρέπει λοιπόν και οι διάφορες σχολές σκέψης των δικαστών να λάβουν υπόψη αυτή τη λογική. Τώρα, ο Λουίς Περέιρα, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστών, θα μας μιλήσει και αυτός για τα θέματα που μας απασχολούν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τις Επιτροπές Ελευθεριών και Νομικών Θεμάτων για την πρόσκληση που μας απευθύνει την τιμή μας να είμαστε εδώ πέρα για να μοιραστώ μαζί σας τις ε, προοπτικές ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης ε, των Δικαστικών. Θα ήθελα να κάνω πρώτα απ' όλα μια εισαγωγή για τον οργανισμό που εκπροσωπώ. Το δίκτυό μας είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός του πολιτικού δικαίου και είναι μάλλον ο μόνος ε, ιδιωτικός οργανισμός που έχει μέλη μόνο δημόσιους φορείς. Και από τα 27 κράτη μέλη, μάλιστα, μαζί με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, που είναι μέλη του δικτύου μας. Έχουμε λοιπόν ως μέλη τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, ε, όπως τη Γερμανία και την Αυστρία, ανώτατα δικαστήρια, όπως αυτό της Κύπρου και της Εστονίας, σχολές δικαστών, υπό την αιγίδα των αντιστοίχων Υπουργείων Δικαιοσύνης, όπως της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, και ανωτάτων και ανώτατα συμβούλια δικαστών όπως στην Ισπανία. Το δίκτυό μας ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια για να αποτελέσει μια πλατφόρμα ανταλλαγής ε, εμπειριών των μελών, των μελών του που είναι υπεύθυνα για την εκπαίδευση 140.000 δικαστών και εισαγγελιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημασία του δικτύου μας αναγνωρίστηκε το 2007 με την ε, απόφαση του δικαστηρίου της, ε, του Συμβουλίου συγχωρείτε, της 12 Φεβρουαρίου του 2007 που αναγνώρισε πως ε, το δίκτυο προωθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευση δικαστών και εισαγγελέων με μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση, συνεισφέρει στην ενίσχυση της αμοιβαία εμπιστοσύνη και βελτιώνει την αλληλοκατανόηση μεταξύ δικαστικών αρχών και διαφορετικών νομικών συστημάτων. Στην ίδια απόφαση του Συμβουλίου αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, πως για να στηριχθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του δικτύου χορηγείται μια πίστοση λειτουργίας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν εκτέλεση αυτής της απόφασης του Συμβουλίου μπορούμε να αναφέρουμε σε εσάς το τι έχει επιτύχει το δίκτυό μας. Το δίκτυο έχει τώρα 45 εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 19 κράτη-μέλη. Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων σημαντική είναι, σημαντικό είναι το πρόγραμμα ανταλλαγής ξεκίνησε το κοινοβουλίο σας. Ξέρετε πως υπάρχουν τρεις βασικές τάσεις ε, όσον αφορά την εκπαίδευση των δικαστών. Έχουμε εκπαίδευση σε μέσα ε, σε ευρωπαϊκό δίκαιο, σε μέσα δικαστικής συνεργασίας, σε ε, γλώσσες και επίσης εκπαίδευση σε ε, διαφορετικά νομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το πρόγραμμα ανταλλαγής εστιάζει ακριβώς σε αυτούς τους τομείς. οργανώσει λοιπόν ένα πρόγραμμα με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο επιτρέπει στους δικαστές, τους εισαγγελείς από κάθε κράτος μέλος να πάνε σε ένα άλλο κράτος μέλος να τους φιλοξενήσει ένας συνάδελφος για να έχουν μία εικόνα για τη λειτουργία του νομικού συστήματος της εν λόγω Επιπλέον, πέρα από αυτό το πρόγραμμα που οργανώσαμε το 2005 έχουμε και άλλους ε, τομείς ε, ανταλλαγών δηλαδή όσα έχουν γίνει σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Eurojust και ε, οργανώσαμε και επισκέψεις για να αποκτήσουν μια σωστή εικόνα της λειτουργίας των οργάνων αυτών οι δικαστές. Για να ανταποκριθούμε δε στα αιτήματα του τομέα αυτού, ζητήσαμε να υπάρξει ένα πρόγραμμα Εράσμους, θα λέγαμε, που απευθύνεται σε νέους δικαστές και εισαγγελείς. Και μπορέσαμε φέτος να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό έργο που απευθύνεται σε αυτό το ειδικό κοινό και μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των μελλοντικών δίκαστων της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίς στη σταδιοδρομία τους. Με το πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία επαφών με τα νομικά συστήματα των χωρών που επισκέπτονται οι νεαροί δικαστές, οι μέλλοντες δικαστές και να μοιραστούν έτσι τις εμπειρίες τους. Μαζί με αυτό έχουμε και άλλα προγράμματα που αφορούν το μίσο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, δηλαδή τα έργα ποινικού δικαίου 1 και 2, μια σειρά σεμιναρίων αστικού δικαίου και ανεξάρτητα σεμινάρια Παράλληλα, ξεκινήσαμε και εκμεταλλευτήκαμε μια δραστηριότητα που υπάρχει εδώ και 8 χρόνια που ξεκίνησε η Πορτογαλική Γερμανική Σχολή Δικαστών ο οργανισμός Θέμης που απευθύνεται σε νέους δικαστές και εισαγγελίες. Και φέτος ε, βλέπουμε πως είχαμε συμμετοχή 42 ομάδων από 23 χώρες. 21, 21 από αυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα είχαμε και άλλα μέσα εκπαιδευτικά, τα γλωσσικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και νέες μεθόδους εκπαίδευσης και έχουμε βέβαια και την λεγόμενη διδακτέα ύλη, δηλαδή κάπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποια μέσα τα οποία θα επιτρέψουν τη γνώση και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτά είναι διαθέσιμα στο σελίδα μας. Ταυτόχρονα Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ε, εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και παράλληλα για να επανέλθω σε αυτό το οποίο έλεγα στην αρχή έχουμε και εκπαίδευση των εκπαιδευτών όπου δημιουργούμε φόρουμ και πλατφόρμες όπου οι εκπαιδευτές από διάφορα κράτη-μέλη μπορούν να μοιραστούν ε, τις ε, μεθοδολογίες που έχουν τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά και την πείρα τους στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Νομολογία. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, θα έλεγα, του δικτύου μας. Έχουμε δικαστές από κράτη-μέλη, κοινέ ευρωπαϊκές αξίες, χρήση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, μια κοινή δικαστική κουλτούρα σε έναν ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο. Για να γίνει αυτό εφαρμόζουμε δύο βασικές έννοιες. Τη μία είναι αποκεντρωμένος σχεδιασμός, θα την έλεγα, και η άλλη είναι αποκεντρωμένη εκτέλεση. Τι σημαίνουν αυτά στην πράξη. Αποκεντρωμένος σχεδιασμός σημαίνει πως αντί να έχουμε να παρέχουμε εμείς στην εκπαίδευση, συλλέγουμε την ε, εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να ορίσουν το πρόγραμμα και να επιλέξουν την μέθοδο με την οποία θα ε, γίνει η εκπαίδευση. Ταυτόχρονα μιλάμε για μια αποκεντρωμένη εκτέλεση που επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να ετηθεί να οργανώσει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα στην επικράτειά του. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο μπορέσαμε να οργανώσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε 19 κράτη-μέλη. Πώς λειτουργούν όλα αυτά. Βεβαίω υπάρχει σοβαρή δέσμευση των μελών και Βεβαίως ε, τώρα μπορούμε να βασιστούμε. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίω είναι η συνέχεια της οικονομική στηριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω συνέχεια, όχι απλά στήριξη. Μάλιστα μπορούμε να λειτουργούμε με την απαραίτητη συνέχεια που απαιτείται στον σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ε, ανάγκες που έχουμε για την περίοδο 2007-2013. Βεβαίως έχουμε ένα ειδικό κοινό ε, και αυτό σημαίνει κάποια πράγματα για τη διαθεσιμότητά τους. Δικαστές και εισαγγελείς δεν μπορούν να σηκωθούν να φύγουν, να αντιλαμβάνεστε από τα δικαστήρια, οπότε πρέπει να γίνεται πάρα πολύ καλός σχεδιασμός. Για να σας δώσω μία ιδέα για το πρόγραμμα ανταλλαγών που ξεκινήσαμε το, θα ξεκινήσουμε το 2014. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Για να ξεκινήσει λοιπόν η πρώτη εισαγωγή του προγράμματος ε, ΕΑΚΟΣ ε, ε, εβδομάδες προγραμματισμού 20 μήνες πριν. Για να επιτρέψουμε λοιπόν και στους συμμετέχοντες ε, και στους φορείς ε, και στις αρχές βεβαίως να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Κάνουμε αυτό ακριβώς ε, τον μακροχρόνιο προγραμματισμό. Και αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε την περίοδο 2014-2020 και η πρότασή μας, ε, δεν τολμάω να το πω έτοιμα, είναι να αφήσουμε τα πράγματα όσο έχουμε. Ο μηχανισμός ε, της χρηματοδότησης ε, λειτουργεί μια χαρά και κατά την άποψή μας κάτι το οποίο λειτουργεί δεν χρειάζεται να το πειράζουμε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την ε, κατάτησή μας, πώς φεύγουμε στους πιο ειδικούς από τα κρατημέλη και ακριβώς εξαρτώμαστε από τα κρατημέλη για τους εκπαιδευτές και επίσης ε, διαδίδουμε, ε, παρέχουμε πληροφορίες από τον τοπό μας και συνδεόμαστε έτσι με αντίστοιχα σε τη μέλη για να μπορέσουμε να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση σε αυτήν την κατάρτιση και εκπαίδευση. Και για αυτόν τον λόγο συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη που έχουν αντίστοιχους φορείς εκπαίδευσης και επίσης έχουμε και στήριξη από την γραμματεία. Για να δούμε τώρα κάποια αριθμητικά στοιχεία. Αρχίζουμε με την ε, ανταλλαγή Φανταζόμαι ότι θα χαρείτε αν σας πω ότι το 2012 είχαμε συμμετοχή 1230 στο πρόγραμμα των ε, ανταλλαγών. Τώρα, όσον ε, αφορά τώρα τις εκδευτικές μας δραστηριότητες, αυτά τα οποία έχουμε οργανώσει στα κράτη-μέλη, φτάσαμε σε ε, κατάρτιση 2.325 δικαστών και εισαγγελίων του 2012. Πάντως ε, αυτός ο αριθμός δεν αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που εξετάζουμε. εδώ βλέπετε, ε, δεν είναι τόσο διάκριτη βέβαια η διαφάνεια, Σα έχουμε μοιράσει την ειδησία έκθεση και τα λέει καλύτερα, φαίνονται καλύτερα και εδώ λέμε ε, τι γίνεται ανά η ημέρα εκπαίδευση. Λέμε εδώ για το τι μαθαίνει κάποιο κάποια μέρα που πέρασε από την εκπαίδευση. Πάντως, δεδομένε αυτέ τι δραστηριότητε, δεν θα πρέπει να θεωρήσει κανεί ότι σταματάει εδώ το βεληνικέ στον γιατί έχουμε και άλλα στα κράτη-μέλη, ε, δραστηριότητε κρατών μελών που χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Και επ' αυτού ε, φτάσαμε του 1937 δικαστέ που μετέσχων με όλου του δυνατού τρόπου. Επομένω, το έχουμε σύνολο 4.350 δικαστών και το 2012. Εδώ βλέπετε σε ένα διάγραμμα την προέλευση αυτών που έλαβαν μέρο μέρος στις μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για τη δραστηριότητα του EJTN. Μας μιλήσατε για το παράδειγμα του Εράσμους για δικαστές. Μίλησατε και για ένα θέμα που συχνά παραμελούμε και που θεωρώ σημαντικό για να δημιουργήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα πρόβλημα της γλώσσας. Γιατί οι δικαστές και οι νομομαθείς είναι οι αριστοκράτες της κουλτούρας. Θεωρούν τη γλώσσα λοιπόν ως ένα σήμαντο εργαλείο. Όχι πολύ σημαντικό πνευματικά. Αυτό είναι λάθος. Χωρίς ε, τη διάδοση μίας κοινής γλώσσας μεγάλη διάδοση μια κοινή γλώσσα δεν πρόκειται να πετύχουμε την οικοδόμηση τη Ευρώπης. Πώς μπορούμε να είμαστε τμήμα μια κοινότητα, όταν δεν καταλαβαίνόμαστε. ένα μιλάει και άλλο δεν καταλαβαίνει. Η Ευρώπη έχει αυτό μεγάλο εμπόδιο. Είναι και πλούτο, αλλά είναι και πρόβλημα παράλληλα. Και αν δεν αντιμετωπίσουμε με ταπεινοφροσύνη και πρακτικότητα αυτό το προδικαστικό ζήτημα, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Δεύτερον, το θέμα της επανακατάρτισης των δασκάλων, της επιστροφής στα θρανία. Και αυτό που είπε ο κύριος Περέιρα για τον πρώιμο σχεδιασμό. Αν θέλουμε να προβούμε στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση των δικαστών, πρέπει να τη σχεδιάσουμε. Και μετά τα αυτά, μπαίνουμε στο θέμα της, του οικονομικού σχεδιασμού. Ο Περέιρα ξέρει ότι ήμουν εισηγητής του για τον κανονισμό που προέβλεπε την ευθετή, τον εφταετό οικονομικό σχεδιασμό για τη δικαιοσύνη, για το τομέα της δικαιοσύνης. Και τώρα που συζητήσαμε και ακούσαμε για το AJTN, φαίνεται πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε και για τα νούμερα που μας δώσατε. Γιατί αυτά που λέγε ο συνάδελφος Ροντβίρεν και αυτά που λέει ο κύριος Περέιρα σε κλείνουν τελικά. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, πάμε στον Εμμανουέλ Κράμπιτ, προϊστάμενο της Γενικής Διάθεσης Δικαιοσύνης. Και το θέμα που επέλεξε είναι να μιλήσει για την κατά αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης που συνδέεται με το πρόβλημα της κατάρτισης και της νομοθεσίας. Δηλαδή, με ποιον τρόπο καταλαβαίνουμε πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο Εμμανουέλ παίρνει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ήρθα εδώ για να κάνουμε αυτό το διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και να μιλήσουμε για ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη. Γιατί πρόκειται για την λειτουργία του δικού τους εθνικού δικαστικού συστήματος. Το κείμενο που παρουσιάστηκε είναι ένα έγγραφο που σκοπό έχει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις ε, εθνικές τους αναμεστάξεις. Υπάρχουν σχετικά έγγραφα και στα, στην άκρη της αίθουσας. Δίνει συγκρίσιμα στοιχεία για διάφορες παραμέτρους που αφορούν τα δικαστικά του συστήματα. Μιλάει για θέματα ανεξαρτησίας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης τους. Γιατί η Κομισιόν αποφάσισε να παρουσιάσει ένα τέτοιο έγγραφο που να μιλάει για τα αποτελέσματα. Γιατί η αποτελεσματικότητα των εθνικών νομικών συστημάτων είναι απαραίτητη για όλη τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ανάπτυξή της. Απαραίτητο γιατί. Γιατί η αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων εξασφαλίζει την υλοποίηση όλων των κανόνων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι τόσο απαραίτητο που είναι και θεμελιώδες δικαίωμα. Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει το άρθρο 47 που λέει ότι όλα τα άτομα του οποίου τα δικαιώματα εγγυάται η εθνική νομοθεσία, όταν αυτά τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί, μπορεί να προσφύγει σε, σε ένα δικαστήριο. Η δυνατότητα αυτή προσφυγής σε ένα δικαστήριο υπάρχει στο σύστημα στην ένωμη τάξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ένα εθνικό δικαστή εφαρμόζει μια οδηγία για την προστασία των καταναλωτών ή για το περιβάλλον, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, για την ενιαία αγορά, ε, λειτουργεί ω Ευρωπαίος δικαστή. Υπάρχει λοιπόν κοινό συμφέρον να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαστικά συστήματα, τα νομικά συστήματα λειτουργούν αποτελεσματικά με ποιοτικό τρόπο για να υλοποιηθούν όλοι αυτοί οι κανόνες που υιοθετήθηκαν εδώ και χρόνια στην, Ιστορική Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, είναι σημαντικό για την αμοιβαία εμπιστοσύνη, για την ανάπτυξη αυτής και για τα εργαλεία συνεργασίες που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό γι' αυτό να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία των εθνικών και τις εθνικές νομοθεσίες, γιατί αυτά θα μας εξασφαλίσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κάτι άλλο αποφασιστικό στην παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας για τον πίνακα αποτελεσμάτων. Αυτό είναι σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη, που όπως ξέρετε είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Και αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το κείμενο, θα επιτρέψει να εμπλουτίσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο που είναι ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Ξάμεινο η μεταρρύθμιση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών είναι μία από τις προτεραιότητες. Η ποιότητα, η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα των δικαστικών συστημάτων της άνομης τάξης των κρατών μελών είναι ένας στόχος που αναφέρεται ρητά στο Ευρωπαϊκό Ξάμεινο. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την προτεραιότητα χρειαζόμαστε συγκρίσιμα στοιχεία και πρέπει να έχουμε συστηματικά πληροφορίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πληροφορίες αντικειμενικές. Σε ορισμένε περιπτώσει αυτό θα μα επιτρέψει να κάνουμε συστάσει ορισμένα κράτη-μέλη, να του επιστήσουμε την προσοχή, να τα ενθαρρύνουμε για να βελτιώσουν τη λειτουργία του δικού του εθνικού συστήματος. Το 2012 έξι κράτη-μέλη έλαβαν σύσταση για τη βελτίωση του δικαστικού του συστήματος. Το 2010 στις 20... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συστάσεις για 10 κράτη-μέλη. Αυτές οι τάσεις μιλούσαν για την ανεξαρτησία μερικές φορές του συστήματός τους, άλλες φορές μιλούσαν για την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητα του συστήματός τους. Ο πίνακα αποτελεσμάτων για την ε, δικαιοσύνη είναι ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε μια βάση για την ανάλυση ανακράτως μέλος που γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του πρώτου πίνακα αποτελεσμάτων του 2013. Καταρχάς, πρέπει να εξηγήσω ότι Ασχοληθήκαμε με τη λειτουργία της ε, πολιτικής δικαιοσύνης, αστικής δικαιοσύνης, ε, αστικό δίκαιο, εμπορικά θέματα, αλλά όχι, δεν ασχοληθήκαμε με την ποινική δικαιοσύνη. Χρησιμοποίησαμε μια σειρά από δείκτες που μπορούμε να τις ομοδοποιήσουμε σε τρεις κατηγορίες. Δείκτες καταρχάς που αφορούν την ε, ταχύτητα των διαδικασιών δικών κτλ. Χρησιμοποιούμε δεδομένα που βγαίνουν από την ε, Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης που επί 10 χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό και που αφορούν τη διάρκεια των διαδικασιών και το ποσοστό υποθέσεων που καθυστερούν, τις εκκρεμείς υποθέσεις κτλ. Ένας δεύτερος αριθμός δικτών που εξετάζουμε είναι δείκτες που αφορούν την ποιότητα. Το να έχουμε δείκτες για την ποιότητα της δικαιοσύνης είναι ένα περίπλοκο θέμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πάρουμε δείκτες για στοιχεία που ενθαρρύνουν την ποιότητα. Και ένα από τα στοιχεία αυτά, ένας από τους δείκτες αυτούς, είναι η κατάρτιση των δικαστών. Θα βρείτε λοιπόν σε αυτό το έγγραφο διάφορες γραφικές παραστάσεις που παρουσιάζουν δεδομένα ε, για στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα, όπως τη χρήση των τεχνολογιών, της πληροφορικής, την κατάρτιση, χρήση της πληροφορικής στη διαχείριση των υποθέσεων του δικαστηρίου. Επίσης έχουμε δείκτες για την ποιότητα που που είναι ας πούμε η μέθοδος αξιολόγησης. Δηλαδή υπάρχουν στα κράτη-μέλη συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης της, δράσης, της δραστηριότητας των ε, δικαστηρίων, ε, δείκτες και στοιχεία για τις, τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Συγγνώμη, και οικονομικούς πόρους. Ένα άλλο στοιχείο που έχουμε είναι δείκτες για, τους, ε, για την εξαρτησία για την αντίληψη που υπάρχει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην εκάστοτε χώρα. Συνειδητοποίησαμε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρούμε δείχτες που να αφορούν την πραγματική διαρθωτική ανεξαρτησία. Αλλά υπάρχουν στοιχεία για την αντίληψη που έχουμε για αυτή την ανεξαρτησία. Και έτσι χρησιμοποίησαμε ένα δείχτη που διαμορφώθηκε από το World Economic Forum και έναν άλλο δείχτη από το World Justice Project που είναι πολύ ενδιαφέροντες γιατί στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η αντίληψη για την εξαρτησία είναι ένα από τα στοιχεία που αναφέρθηκε και από το ίδιο δικαστήριο αλλά και από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Si vous Αν ε, φιλομετρήσετε το έγγραφο, είναι δύσκολο να πείτε ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής ή ποιος είναι ο σκράπας. Επίτηδες το κάναμε αυτό. Γιατί ο σκοπός αυτού του πίνακα δεν είναι να κάνουμε καλυστία, ούτε να βάλουμε βαθμούς για να πούμε «Να, εσύ είσαι ο καλύτερος, είσαι ο κακός μαθητής». Πρέπει να έχουμε πάρα πολύ, πολλές αποχρώσεις στην ερμηνεία, γιατί κάποια χώρα μπορεί, ας πούμε, να έχει πολύ καλά νούμερα για τη διάρκεια των αστικών υποθέσεων πονδικών για αστικές υποθέσεις, αλλά πολύ κακή για διοικητικέ υποθέσεις. Μία χώρα μπορεί να χρησιμοποιεί πολύ τις νέες τεχνολογίες, αλλά μην είναι πολύ καλή, ας πούμε, σε θέματα διεκπαιρέωσης των εκκρεμών υποθέσεων. Επομένως, υπάρχουν πολλές αποχρώσεις πίσω από τα γραφήματα και αυτό δείχνει την περιπλοκότητα του εγχειρήματο το να παρουσιάσουμε υπομορφή πίνακα την ε, επίδοση των διαφόρων συστημάτων. Όσον αφορά τώρα τη διάρκεια των διαδικασιών υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Το βλέπετε αυτό σε όλες τα γραφήματα και βλέπετε το εν τρίτον των μελών έχουν μια διάρκεια των διαδικασιών που είναι δύο φορές πιο μεγάλη από ότι η πλειοψηφία των κρατών μέλων. Τώρα όσον αφορά τις ε, τεχνολογίες κατάρτισης και εδώ έχουμε μεγάλη ανισότητα. Πολλές φορές τα πράγματα είναι περίπλοκα. Μπορεί να έχουμε μια χώρα που έχει πάρα πολύ καλές παραμέτρους όσον αφορά την χρησιμοποίηση τεχνολογιών για τη διαχείριση των δικαστηρίων, αλλά δεν έχει καλές επιδόσεις όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών για τις σχέσεις με τους διαδίκους ή τους δικηγόρους. Οπότε και εν προκειμένου Έχουμε αυτά τα γραφήματα τα οποία μας δείχνουν μεγάλη ανισότητα. Βεβαίω. Δεν σημαίνουν αυτά ότι μπορούμε να εξαγάγουμε αυτομάτως κάποια συμπεράσματα. Θα πρέπει να μας διακρίνει ταπεινότης όταν ερμηνεύουμε αυτές τις παραμέτρους. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να πάει κανείς παραπέρα. Όταν θα κάποια κράτη-μέλη έχουν σωρεύσει κακές επιδόσεις όσον αφορά πολλούς, πολλούς, πολλές προγραμμές, πολλά κριτήρια, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι κρύβει από αυτό. Οπότε για άλλη μια φορά αυτό είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο να βοηθήσει τα κρατημέλη να έχουν μια οπτική συγκριτική και να εμβαθύνουμε όσον αφορά τους ε, διαφορετικούς λόγους που κρύβονται πίσω από κάποιες επιδόσεις που δεν εμφανίζονται και τόσο άριστες. Τώρα για την Επιτροπή, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε ένα διάλογο με τα κράτη-μέλη και μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε σε κατανόηση και μπορούμε έτσι να προβούμε σε συστάσεις για το μέλλον. Αυτός ο χάρτης επιδόσεων έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και σε σχέση με το τι τομείς καλύπτονται. Είπαμε στην αρχή ότι έχουμε αστικές, ε, εμπορικές και δυτικές υποθέσεις που καλύπτονται. Και είναι εξελικτικό όμως και για τους δείκτες. Και όπως σας έλεγα είναι το θέμα της ανεξαρτησίας, όπου εκεί τα πράγματα επιδέχονται βελτίωση. Και είπαμε ότι αυτό να το κάνουμε με τα δίκτυα με τα ανώτερα δικαστήρια, γιατί υπάρχουν πολλά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έργο το οποίο θα το κάνουμε για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πληροφορίες όσον αφορά την δομική, διαρθρωτική ανεξαρτησία των δικαστικών νομικών συστημάτων, επίσης και επιτόπου μελέτες. Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία είναι μέση όρη, μαθηματική αλλά επί τόπου θα καταλάβουμε ε, στη λεπτομέρεια το τι ισχύει και τι προβλήματα σοβούν ή στην, στη λειτουργία των δικαστηρίων είναι κατακλείδη τώρα. Θέλω να σας πω το εξή. Παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αυτή την πρωτοβουλία το ότι έτσι εκφράζεται η βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταλάβει καλύτερα τι συμβαίνει επί τόπου. Επί μικρόφωνικο διάστημα εμείς όλα τα θεσμικά όργανα ε, ασχολούμεθα με το να παράγουμε κανόνες δικαίου. Τώρα όμως με τέτοια προσπάθειες προσπαθούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται στην πραγματικότητα. Να, ποια είναι η διαφορά. Του τι λέμε εδώ από τις Βρυξέλλες και τι επιζητούν, τι προσδοκούν οι Ευρωπαίοι. Επενδύσαμε λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια. Με όλους τους εμπλεκομένους και ενδιαφερομένους. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη. Και ακριβώς όπως και το θέμα της κατάρτισης των δικαστών, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επισέλθουμε στην ε, πολυπλοκότητα της εφαρμογής του κοινωνικού δικαίου. Και σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για την εισήγησή σας. κύριε Κράμπη. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα του δίκτυ, του, του, του φύλου επιδόσεων ήταν εξαιρετική ιδέα. Το να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει επί τόπου, στην πράξη, στην κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, για να μην πω απαραίτητο. Να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία, πληροφορίες χρήσιμες, το να δούμε κατά πόσο υπάρχει ποιότητα, αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στη δημοκρατική Ευρώπη πρέπει να ομολογήσουμε όμως υπάρχουν μερικές χώρες με πρόβλημα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Είναι πολύ λεπτό θέμα και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρενέβη για να καταδείξει το πρόβλημα της Ουγγαρίας. Λυπάμαι, αλλά οφείλω να το πω αυτό. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν προβλήματα ανεξαρτησία στη χώρα αυτή. Και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ακούστηκαν. Για την ποιότητα των ιδεών που κυκλοφορούν, το κατά πόσον διαδίδονται καινούριε ιδέες, κατά πόσον υπάρχει η έννοια της αυτοκατάρτισης στον χώρο και τον κόσμο των δικαστών. Όλα αυτά είναι αντικειμενικά θέμα, ε, στοιχεία, θέματα. Ε, η διάρκεια, ας πούμε, των διαδικασιών είναι πολύ σημαντικό θέμα και αντικειμενικό. Και αυτό το ερώτημα θέλω να θέσω στον κύριο Κράμπιτ. Πέρα από αυτές τις τρεις παραμέτρους, που είναι σίγουρα οι πιο σημαντικές. Αλλά το ερώτημα που θέσαμε στον εαυτό μας αυτούς τους τελευταίους μήνες είναι ότι από την αξιολόγηση των του προγράμματο τη ε, Στοκχόλμης, οι τρει αρμόδιες κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, ΛΥΜΠΕ, ΑΦΚΟ και ΓΙΟΥΡΙ, ε, προετοιμάζουν μια κοινή σύνοδο, μια συνεδρίαση κοινή τον Ιούλιο για να συζητήσουν τα θέματα δυσκολίες εφαρμογής. Μερικές φορές ε, το πρόβλημα έγκυται στη φύση των κανόνων που παράγουμε. Παρά τη μελέτη αντικτύπου, προωθούμε νομοθετήματα θεωρώντας ότι θα έχουν το χι αποτέλεσμα, παραβλέποντας τις πραγματικές απτές δυσκολίες παραβλέποντας τη φύση της κοινωνίας στην οποία παρεμβαίνουμε με το νομοθέτημα αυτό. Έχουμε λοιπόν έτσι μια αφηρημένη εικόνα της πραγματικότητας. Ο πίνακας αυτός αποτελεσμάτων θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμος αν βάλουμε και άλλες παραμέτρους. Είναι... Πρέπει, Το πρόγραμμα προβλέπει τις παρεμβάσεις των εθνικών ε, βουλευτών. Έχω τρεις εθνικούς, εθνικούς βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Και για να μην ε, ξεπεράσουμε το χρόνο μας, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, Ρικάρντο Ροντρίγκε που εκπροσωπεί την Πορτογαλική Βουλή. Τώρα, εάν όσο μιλάει ο κύριος Ροντρίγκε θέλει και κάποιο άλλο βουλευτή να πάρει το λόγο, να μα το πει. Ρικάρντο Ο κύριος Ρικάρντο Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά βρισκόμαι εδώ σε αυτή τη συνάντηση του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Έτσι αποκτούμε εμπειρία όσον αφορά την εξέλιξη του δικτύου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ε, συζήτηση αυτή για την ε, δικαστική ευρωπαϊκή κουλτούρα. Είναι βέβαια εδώ το ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων. Φτιάξαμε την κοινή αγορά, η οποία έχει συνέπειες όσον αφορά την εξέλιξη και την διαμόρφωση του δικαίου. Κάθε χώρα θα πρέπει να παραγάγει την νομοθεσία της. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης κάνει το ίδιο. Όμως η πολυνομία φέρνει προβλήματα εφαρμογής του δικαίου. Ακούσαμε τα της κατάρτισης γιατί ένα άλλο ζήτημα είναι και οι νομικοί, το τι θα κάνουν αυτοί, δηλαδή που κάθε μέρα ασχολούνται με τα δικαστήρια, εκτός δικαστές λοιπόν, είναι οι δικηγόροι που υπεστούν τους ε, πελάτες τους, αλλά και το θέμα της πληροφόρησης του κόσμου για τους νόμους. Άρα, χρειάζεται συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση όπως αναφέρθηκε. Δεν νοείται το να έχουμε καλούς δικαστές και καλούς δικηγόρους αν εκείνοι δεν περνάνε από αυτήν την συνεχή εκπαίδευση. Και όπως είπαμε, θα πρέπει να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο η οργάνωση αυτής της εκπαίδευσης. Και θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση κάποιοι εκπαιδευτές να κάνουν αυτή την εκπαίδευση. Να μην φτάνουμε στο σημείο να έχουμε αντιφατικές αποφάσεις στο δικαστήριο. Επίσης, για τους Ευρωπαίους, είναι απαράδεκτες και αυτές οι δικαστικές αποφάσεις. Πράγματι για μας, παράκτες για τους Ευρωπαίους, άρα θα πρέπει μέσω της εκπαίδευσης να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Και αντίστοιχα θα πρέπει να γίνει η διαμόρφωση της νοοτροπίας, της σκέψης των νομικών. Πολύ σημαντικά αυτά για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Έχω μια ιδέα, μια πρόταση. Άκουσα τι είπε ο κύριος Λουίς Περέιρα. τύπωσε κάποιους προβληματισμούς για την επαγγελματική κατάρτιση. Βέβαια, ο πρόεδρος τόνισε ότι υπάρχει πρικοδότηση που προβλέπεται για την εκπαίδευση. Πάντως προβληματιζόμαστε γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης και οι πολίτες να μπορούν να απευθυνθούν σε έναν δικηγόρο. Όμως και ο δικαστής και ο δικηγόρος υποχρεούνται να είναι ενημερωμένος. Και αυτό επομένω κάνει η εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν έχω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. <laughs> Θα απαντήσω στην τελευταία μόνο παρατήρηση, γιατί κατάλαβα ότι με αφορούσε. Ε, προς εμένα απευθυνόταν, γιατί είμαι ο εισηγητής. Δεν αποφασίζω εγώ, εισηγητής είμαι. Η πρόταση για συμμετοχή του EGTN στο 7 πρόγραμμα έχει γίνει δεκτή. Φυσικά δεν έχουμε ολοκληρώσει συζήτηση για τον προπολογισμό και επομένω δεν ξέρουμε τα τελικά ποσά που θα πάρει κάθε τομέα. Δεν ξέρω ε, τι χρήματα θα πάνε για τον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι ακόμα υπό συζήτηση το θέμα, αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα για κονδύλια στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. θα παρουσιαστούν τα αιτήματα και θα τα εξετάσουμε με βάση τους κανόνες. Επομένως, θα δούμε τώρα στην πράξη θα γίνει. Ο Μίσα Σεβερίνσκι ζητάει το λόγο τώρα. Είναι Πολωνός βουλευτής. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από τον τίτλο της συζήτησης αυτής, του πάνελ αυτού και από μια σειρά από ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, κατάλαβα ότι μιλάμε, ότι μιλάμε για την αποτελεσματικότητα της δικαστικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Θα ήθελα να κάνω και μια αξιολογική κρίση για αυτήν την κουλτούρα. Είμαι καθηγητής νομικής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ως τέτοιος δεν θέλω ότι υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή κουλτούρα για τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν κοινά θεμέλια για την, τον τρόπο που λαμβανόμαστε εμείς στην Ευρώπη το δίκαιο. Ίσως είναι, σας φανεί υπερβολική αυτή η δήλωση, αλλά νομίζω ότι είναι αληθής. Ας χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό, τον σημερινό ορισμό ε, που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νομοθέτη σήμερα στην Ευρώπη ή δικαστής. Ε, τον ορισμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ανθρώπινη ελευθερία, την ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι ερμηνείες, ή μάλλον αυτοί οι ορισμοί διαφέρουν. Ρωτήστε. Τους μεν και τους δε. Πότε αρχίζει η ζωή θέσετε ερωτήματα για την άμβλωση, για την ευθανασία, για τη διαδικασία in vitro, την τεχνική γονιμοποίηση. Για όταν ζητάμε άδειες να κάνουμε πειράματα με ανθρώπινα και ζωικά έμβρια. Οι γνώμες διαφέρουν, οι ορισμοί που χρησιμοποιεί ο καθένας διαφέρει. Ο καθένας χρησιμοποιεί διαφορετικές έννοιες, ακόμα και, μια, και κάποιες κλασικές έννοιες, όπως η περιουσία, η κυριαρχία. Δεν τις ερμηνεύουμε, δεν τις αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μιλάμε για ουσιώδεις ορισμούς. Κι όμως η ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα τις αντιλαμβάνεται, δεν είναι μία, είναι κατακαιρματισμένη για να μην πω στρεβλωμένη. Τώρα, για τις εξελίξεις αυτής της ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας, για την πρόοδό της. Μην ξεχνάτε ότι οι φορείς αυτής της ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας είναι άνθρωποι και δεν είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τυφλά τον νόμο. Ερμηνεύουν τον νόμο. Την εφαρμόζουν απλώς. Τον εφαρμόζουν τον νόμο. Αυτά ευχαριστώ. Caro collega, io Αγαπητοί, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να εκφράσω την άποψή μου και εγώ με τη σειρά μου, γιατί θέσατε πολύ σημαντικά προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε στην Ευρώπη υπήρχε η δουλοπαρικία. Κάποτε υπήρχε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της ανθρωπότητας, ο Αριστοτέλης, που θεωρούσε ότι η έννοια των σκλάβων ήταν κάτι το σωστό και το δίκαιο. Αν είχαμε την ίδια νομική κουλτούρα με την εποχή του Αριστοτέλη, ε, θα είχαμε την... σήμερα θα επιτρέπαμε τη δουλεία. Κάποτε το φέουδο ήταν η βάση της κοινωνίας. Αλλά μετά κάποια στιγμή όλοι οι πολίτες απέκτησαν την αρχή της ισονομίας. Αυτό ξεκίνησε με τη Γαλλική Επανάσταση ή με το, με το χαμπέους κόρπους. κόρπους. Ναι. Αυτά την εποχή του Μεσαίωνα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν δύο αρχές, δύο εξουσίες. Και μετά το μοντέρνο κράτος δημιούργησε την έννοια της ε, κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας, η οποία εν συνεχεία θεωρήσαμε ότι ανήκει στο λαό. Επομένως, διάφορες ε, από αυτές τις θεμελιώδεις έννοιες αλλάζουν, όπως αλλάζει και η ιστορία. Και εμείς ανήκουμε σε μια ιστορική στιγμή η οποία επλήγει από ένα κυκλώνα. που διαμορφώθηκε από την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, δημιουργήθηκε η έννοια της ευρωπαϊκής κοινότητας, που είναι μια ιδέα εντυπωσιακή. Οι μελετητές του διοικητικού ε, δικαίου λέγανε ότι δεν υπάρχει διοίκηση χωρίς κράτος. Και εμείς έχουμε μια διοίκηση στην Ευρώπη χωρίς να έχουμε κράτος. Και δεν θέλουμε να έχουμε ένα τέτοιο κράτος. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, θέλουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έννοιες αλλάζουν, εξελίσσονται. Και η γοητεία τους είναι ότι εμείς βρισκόμαστε και ζούμε σε αυτό το χωνευτήρι. Υπάρχουν ιδέες του παρελθόντος που ε, επιβιώνουν και υπάρχουν και νέες ιδέες. Και το πρόβλημα είναι ότι η δημοκρατία στην Ένωση οδηγεί στην ορίμαση και κάποιων αρχών. Και οι αρχές αυτές μετά διαδίδονται και τις μοιράζονται όλοι. Αυτή είναι η φτωχή και ταπεινή γνώμη ενός ε, ομολόγου σα, ενό άλλου δικαστή νομική, ε, ε, καθηγητή νομικής. Νομίζω όμω ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα, να δούμε και αυτή τη γοητεία που έχει η καινοτομία. Εξού και η συζήτηση που κάναμε σήμερα. Ότι όταν συγχωνεύουμε, όταν παντρεύουμε διαφορετικά πράγματα, δημιουργούνται καινοτομίες. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Φυσικά δεν μπορώ να σας απαντήσω σε όλα με τις ε, φτωχές και ταπεινές μου τα απαντήσεις, αλλά προσπάθησα. Ε, θα δώσω το λόγο στον Ανδρέας Μαπουρίρες, αν πρόφερα καλά το όνομά του. Μάλλον δεν το πρόφερα καλά. Από την Κύπρο. Μια χαρά το είπατε κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για τη δική μου εμπειρία όταν το 1981 πήρα την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Το σοκ που είχαμε οι δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα από τότε μέχρι σήμερα ήταν μεγάλο. Ανατράπηκαν όλα όσα μάθαμε στο Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 70. Μπήκαμε σε ένα εντελώς καινούριο περιβάλλον ζήσαμε τη σταδιακή ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιδέας και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα φτάσαμε να μιλάμε για συνένωση των δικαίων, αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, ενιαία όργανα και θεσμούς. Εκείνοι που μπορούν να αφομοιώσουν καλύτερα τα δεδομένα αυτά είναι οι νέοι. Όπως συμβαίνει στη χώρα μου, έτσι και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα του δικηγόρου, οι νέοι θα πρέπει να ασκηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα δικηγόρο και να δώσουν εξετάσεις. Θα πρέπει να δοθούν οδηγίες σε όλα τα κράτη να περιλάβουν θέματα ευρωπαϊκού δικαίου στην εξέταση, στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Εμείς μάθαμε ό,τι μάθαμε και διαβάζουμε τα βράδια για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε το νέο νομικό περιβάλλον. Δεν θα ξεχάσω τη σύγχυση που είχαμε όταν μετά το 2004 η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δικηγόροι προσπαθούσαν να καταλάβουν, να αντιληφθούν την έννοια του προκατακτικού ερωτήματος του άρθρου 234 τώρα 267 έβαζαν ερωτήματα και είχαν την απέτηση να εξεταστούν προκατακτικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αυτά να εμπίπτουν στην έννοια του preliminary question, του προκατακτικού ερωτήματος εκπαίδευση τόσο των δικηγόρων όσο και των δικαστών είναι διαβίου. Εκεί που πρέπει να δώσουμε όμως μεγαλύτερη έμφαση είναι στους νέους δικηγόρους και στους νέους δικαστές. Γιατί εκείνοι είναι πιο προσαρμοσμένοι και στη ψηφιακή τεχνολογία και στους νέους θεσμούς γιατί αυτοί θα τους δουλέψουν και θα τους αναπτύξουν την 20 ετία που μας έρχεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαπουρίδη, για την παρουσίασή σας, για τα σχόλιά σας, γιατί μπορώ να πω ότι συμφωνώ απόλυτα ότι σε αυτή την ιδέα της εξέλιξης της επαγγελματικής ζωής, οι δικηγόροι, οι δικαστές, πρέπει να έχουν υπόψη τους και να μην ξεχάνε ποτέ τους καινούριου δικαστές που μόλις πέρασαν ένα διαγωνισμό. Εντάξει, το βρετανικό σύστημα είναι λίγο διαφορετικό, αλλά του καινούριους δικαστέ, λοιπόν που μπαίνουν τώρα. Γίνονται δικαστέ και όμω δεν σταματάει ποτέ αυτή η ιστορία, τα, οι διαγωνισμοί, μια ολόκληρη ζωή συνεχίζουν να καταρτίζονται. Διαβίου μάθηση λοιπόν. Και τώρα τελευταίος βουλευτής είναι ο Βίτο Κρίμη, ο οποίος είναι συντοπίτης μου Ιταλός, θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την Ιταλική εμπειρία, έτσι, εν είδη παραδείγματος. Ο κύριος Μπερλίνγκο φυσικά τη γνωρίζει την Ιταλική πραγματικότητα. Έχουμε το Ανώτο, Συμβούλιο της, το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και, που έχει δημιουργήσει και μία σχολή πρόσφατα. Υπάρχουν και αποκεντρωμένα κέντρα. Δηλαδή, υπάρχουν δικαστές ε, που στέλνονται σε κατατόπους, πούμε, για την αποκεντρωμένη κατάρτιση. Την τελευταία χρονιά των σπουδών ε, στέλνουμε και ειδικού για ευρωπαϊκά θέματα είτε κάποιο ασχολείται με το ποινικό δίκαιο, είτε με το αστικό δίκαιο. Μαθαίνει δηλαδή την, το ευρωπαϊκό ποινικό σύστημα, ας πούμε, και το ευρωπαϊκό αστικό σύστημα. Τώρα, αυτοί που πλαισιώνουν τους δικαστές για να τους βοηθήσουν, ας πούμε, το κάνουν μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό, αλλά ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός. Δεν αρκούν τα άτομα αυτά. Νομίζω και σα μιλάω πάντα για την Ιταλία, έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ότι μπορεί να ισχύει και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να βρούμε μηχανισμού. αξιολόγησης της κατάρτισης κατά τη διάρκεια της καριέρας ενός δικαστή. Ειδικά το, το πόσο καταρτίζεται σε ευρωπαϊκά θέματα. Ακούσαμε όλα αυτά περί δικτύων, ε, περί ανταλλαγών ε, εμπειριών των ε, δικαστών των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε την εξή διάκριση. Καταρχάς, εντάξει, υπάρχει το επίπεδο της καθημερινότητας των δικαστών. Αυτό που λείπει όμως στην Ευρώπη είναι ότι αυτό που δεν ε, υπάρχει είναι η άμεση γνώση της δικαιοσύνης από τον απλό πολίτη. Είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να βάζει κάποιο λέξη κλειδιά στο Google και να βγαίνουν κάποια πράγματα σοβαρά που θα έχουν ελεγχθεί από δικαστές ούτω ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να συνειδητοποιεί ποια είναι τα δικαιώματά του. Μιλάω βέβαια για την εξοικείωσή του με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι, για αυτά που είπε τώρα ο Πολωνός ε, βουλευτής, πέρα από τα όσα είπε ο κύριος Μπερλίνγκουερ με τα οποία συμφωνώ, θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω κάποια πράγματα. Μίλησε για κάτι πολύ σημαντικό, ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας βασικές έννοιες με τελείως διαφορετικό τρόπο στην Ευρώπη. είπατε ότι δεν υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη για βασικές έννοιες. Αλλά κοιτάξτε, πλησιάζουμε. Σήμερα είμαστε πολύ πιο κοντά από ό,τι χρόνια πριν. Είναι μια διαδικασία. Είναι μια πορεία που πρέπει να γίνει. Και για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, καταρχάς θα πρέπει να σταθούμε στην ε, σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση ε, καλών δικαστών και δικηγόρων στην Ευρώπη. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν αρκεί μόνο αυτό, να έχουμε και στις τις σωστές ε, αρχές για την εφαρμογή του δικαίου. Να δούμε δηλαδή πώς εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο σε κάθε χώρα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οικονομική ένωση, αλλά είναι και ένωση δικαίων. Ευχαριστώ κύριε Κρίμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίως για αυτό που είπατε για την αποκεντρωμένη κατάρτιση και για το ότι πρέπει να γίνει αυτή η κατάρτιση υποχρεωτική. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ιταλίας, θέλω να πω, ενέκρινε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται European Gaius, ε, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της Εουρίνφρα το παράδειγμα αυτό που ακούσαμε για την Ορλανδία, του δικτύου αυτού που μας παρουσίασε ο κύριος Βίντερ στην πρώτη παρέμβαση. Ευνευστήκαμε λοιπόν από αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Ένα από τα πράγματα που υπόθηκε που μου έμεινε είναι αυτή η έννοια ότι το να φτιάξουμε μια ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα δεν σημαίνει ότι εντάξει φτιάχνουμε καλούς επαγγελματίες μόνο, κάτι που είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να διαμορφώσουμε και τους πολίτες μας. Πρέπει να διαμορφώσουμε και να εγγράψουμε στο μυαλό των πολιτών και την ιδέα της ευρωπαϊκής ηθαγένεια. Γιατί πιστεύω ότι μία από τις δυσκολίε εφαρμογή, ένα από του λόγου, της δύσκολης εφαρμογής που δεν μπορεί να τον ανακαλύψει το scoreboard είναι το γεγονός ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι πλεονεκτήματα έχουν τα οποία απορρέουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έχουν ιδέα για τα δικαιώματά τους, δεν τα ξέρουν. Και επομένως δεν ενδιαφέρονται. Και μόνο μια σωστή προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει πριν ακόμα καταρτήσουμε σωστά τους δικαστές. Υπάρχει το θέμα των πολιτών λοιπόν. Αυτό το θέμα αφορά το λαό δηλαδή, τους ευρωπαϊκούς λαούς τέλος πάντων. Αυτό που είπε λοιπόν ο κύριος Κρίμη είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω τους ομιλητές αν επιθυμούν να απαντήσουν με δύο λόγια. αν το επιθυμούν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι δικότες μου είναι οι πληροφορίες, η πληροφόρηση, η προσβασιμότητα στο κοινωνικό δίκαιο και μεγάλη μεγάλη μου χαρά σε αυτές τις σκέψεις για το πώς το κοινωτικό δίκαιο θα είναι προσβάσιμο ε, και στους πολίτες. Για το κοινωτικό δίκαιο Εντάξει, είναι η δουλειά των επαγγελματιών, αλλά είναι φτιαγμένο και για τους Ευρωπαίους οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να ωφελούνται από αυτό. Και έχω να προσθέσω στο το ότι η κατάσταση δεν είναι και τόσο ε, δυσάρεστη. Γιατί το κοινωτικό δίκαιο εφαρμόζεται από τους εθνικούς δικαστές γιατί έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο. 80% των υποθέσεων. Επομένω, ακόμα και αν το ξέρει ο εθνικό δικαστή, εφαρμόζει το κοινωτικό δίκαιο. Βεβαίω υπάρχει αυτό το, το, το, το περιθώριο, ε, αυτή, αυτό το παραπάνω, όπου πρέπει να κινηθεί κάποιος ειδικό και τότε ωφελείται κανείς, εάν ε, έχει ε, την, την ειδική γνώση και ωφελείται αν εφαρμόσει το κοινωτικό δίκαιο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι προσβάσιμο το κοινωτικό δίκαιο και όπως είπα στην εισηγησή μου αυτή η ηλεκτρονική πύλη θα πρέπει να είναι ε, ηλεκτρονική πύλη που να μπορούν να, να, να, να, να την χρησιμοποιούν και οι πολίτες. Ο κύριος Περέιρα. Ναι. Επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου. Η ehm, μου γλώσσα να σας πω δύο λόγια για το μέλλον της πληροφορίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρμοδιότητα όλων των μερών και την αναγκαιότητα του να υπάρχει συνεχής επικαιροποίηση, ενημέρωση. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι το μυαλό μας είναι σαν ένας σκληρός δίσκος των 5 MB. Δηλαδή, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι οι βασικές γνώσεις να διαβιβάζονται. Οι βασικές γνώσεις που επιτρέπουν την κατανόηση του νόμου, του δικαίου. και θα πρέπει κανείς να ξέρει πώς θα προσαρμόσει τις δυνατότητές του σε ό,τι επιβάλλεται να κάνει. Από πλευράς τώρα διεθνούς ε, δικαίου, πλώς του τι γίνεται διεθνώς, σύμφωνα σε αυτό που είπε ο κ. Μπαρλιγκουέρ για την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και συμφωνώ και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φαντάζομαι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να αλλάξει την τοποθετησή της για να προσαρμοστεί στα όσα θέλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτή την δικαστική κουλτούρα την ευρωπαϊκή. Εδώ είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί όσον αφορά ε, τον ορισμό, τον ορισμό των ενιών. είναι δικαστική κουλτούρα θα πρέπει καταρχήν να είναι κάτι σύνομο, όμως από την άλλη μεριά το περιεχόμενο του νόμου ε, συνήθως περιέχει και ε, στοιχεία διοντολογικά, ηθικά, ε, στοιχεία από τις ενωμένες τάξεις. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποιες αξίες που είναι σε πάρα πολύ ψηλό βαθμό κοινέ. Όταν επομένω έρθει η ώρα εφαρμογής του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια μιας κοινή δικαστικής ε, κουλτούρας ε, και νοοτροπίας που τελικά είναι η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Πρόεδρε, έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για να καλύψουμε ό,τι χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο πίνακας επιδόσεων λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατές υπάρχουσες σχέσεις. Ωραία, είναι πολύ σημαντική η αξιολόγηση της νομοθεσίας, αλλά για πρώτη φορά έχουμε ένα σύστημα που έχει τέτοια προσέγγιση το να αξιολογεί τη λειτουργία ολόκληρου του εθνικού συστήματος. και εξετάζονται και διαφορετικά νομοθετήματα. Οι οδηγίες, οι κανονισμοί, η αξιολόγηση επομένω του νομοθετήματος είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ο βασικός στόχος. Πάντως πέραν αυτού, αν κάτσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα πώς το σύστημα δικαιοσύνης λειτουργεί, τότε μπορούμε να βρούμε και άλλες παραμέτρους και άλλα κριτήρια. γιατί μιλούμε τώρα και για την υποχρεωτική κατάρτιση των δικαστών. Θα ήταν πάντω ενδιαφέρον να ξέρουμε τι γίνεται με την μη υποχρεωτική κατάρτιση των δικαστών. Τελευταία παρατήρηση τώρα όσον αφορά του διαφορετικού ορισμού. Είναι σαφέ. Όταν θέλουμε να έχουμε συγκριτικές πληροφορίες για το εθνικό σύστημα δικαιοσύνης είναι πω αυτό είναι τόσο διαφορετικό τόσο διαφορετικό και σχετικά τέτοια λέμε. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής. Επομένως, εάν λάβετε υπόψη το τι ισχύει, τη δικονομία έχει κάθε χώρα, τότε και από εκεί μπορεί να βρείτε κάποια κριτήρια. Φυσικά θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ την ερμηνεία των δεδομένων, αλλά πάντοτε μπορεί κανείς να βρει τον κοινό παρονομαστή και έτσι να μπορεί να κάνει τη σύγκριση αλλά να είναι πάντοτε, πάντοτε προσεκτικός όσον αφορά τον, τον, την ερμηνεία. Οι δείκτες αυτοί, τα κριτήρια αυτά, αφορούν κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Αντίληψη, ενεξαρτησίες, διάρκεια, ε, κατάρτιση δικαστών, πέραν των ιδιομορφιών κάθε δικαϊκού συστήματος. Πάντοτε υπάρχει και κοινός προνομαστής. Όχι, δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα για όλους. Φυσικά και σεβόμαστε τη νομική παράδοση του καθενός. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε και να σεβαστούμε την κουλτούρα, την νομική. Και έτσι να προχωρήσουμε με νομική δημιουργικότητα. Ευχαριστώ. Να σας πω προσωπικά θεωρώ ότι η συνάντηση ήταν πάρα πολύ θετική και πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους τρεις που είστε τώρα εδώ στο πάνελ και που έχετε συμβάλει σε αυτό το οποίο λέμε. Νομίζω ότι τώρα διαμορφώσαμε μια ιδέα για το τι ισχύει για την ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα. Να ευχαριστήσω και τους ελληνικούς βουλευτές. Τώρα όμως θέλω να δώσω τη σκητάλη στον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών το λόγο. Τον καθηγητή Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστώ όλους και όλες. Για να κλείσουμε αυτή την μακρά διακοινοβουλευτική διάσκεψη ε, πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθαν ε, στα πάνελ και το πρωί. Από Europol, ε, σύμφωνα με τη συνέχεια της Λισαβόνας, αυτούς που μας μίλησαν για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, τη συνεργασία στα θέματα ποινικής δικαιοσύνης, για την προσέγγιση των διαφορετικών εθνικών ποινικών δικαίων είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλο ένα και πιο σημαντικό. Θα πρέπει να μην το ξεχνούμε. Μην ξεχνούμε ποια είναι η πραγματική σημασία αυτού του γεγονότος. Γιατί ακριβώς ήταν ένας από τους λόγους μας έκαναν να συγκαλέσουμε τη σημερινή συνάντηση. για το χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης, αλλά είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο κομμάτι της ημερίδας μας και της συζήτησης. Γιατί διαχρονικά η Ευρώπη έχει δει, γίνει μάρτυρας κατακτήσεων, αιματοχυσίας, εθνικισμών εμφυλίων πολέμων. Όλα αυτά στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Παντού. Και επανειλημμένα. Όμως, τελικά, βρέθηκε κάτι το οποίο λειτουργεί και αποδίδει σε αυτό το επίπεδο. Είναι το δίκαιο. Ας το κάνουμε δημοκρατικά όμως, ας το δούμε δημοκρατικά, να εμπλέξουμε να φέρουμε κοντά σε αυτό το κοινωτικό δίκαιο τους πολίτες και να συνδυαστεί επομένω ε, σε βορμός προς τον νόμο με την ικανοποίηση από αυτόν. Οπότε να εμπλακούν και οι επαγγελματίες νομικοί, φυσικά και οι δικαστές και οι εισαγγελίες από όλα τα κράτη-μέλη. να τους εμπλέξουμε. Γιατί νομίζω ότι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της ημερίδας μας αυτούς καλύψαμε. Και αυτό άλλωστε και προς το δικό τους συμφέρον. Έχουμε και την πολιτική διάσταση. Πρόκειται για συνταγματική φιλοδοξία του χώρου δικαιοσύνης ελευθερίας κλπ. Να, τι είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ότι θα πρέπει, η νομική μας κουλτούρα θα πρέπει να καλύψει τους γλωσσικούς φραγμούς. Κάθε είδους δυσκολίες. Ένα σωρό τεχνικού, τεχνοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια. Γιατί υπάρχει πολυμορφία σε Ευρωπαϊκή και δεν είναι θέμα οικογενειών ενόμων τάξεων, υπηρετικό, αγγλοσαξονικό δίκαιο. Καμία ενόμη τάξη δεν μοιάζει με άλλη στην Ευρώπη. Οπότε θα πρέπει τόσο από τα τεχνικά προβλήματα να ξεπεράσουμε και την πολιτική αβουλία που υπάρχει ούτως ώστε να έχουμε κάποια κοινά νομικά εργαλεία. Όμως αυτό πρέπει να γίνει αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Θα συνεργαστούν χέρι-χέρι τα εθνικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, αυθεντικά ευρωπαϊκό. Και έτσι αυτές τις νομικές παραμέτρους να τις υιοθετήσουν οι δικαστές κάθε κράτος μέλους. Και έτσι να υπάρχει ένα πραγματικά ε, μια πραγματικά ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα με βέβαια πρωταγωνιστή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και για τα ποινικά ζητήματα και να έχουμε επίσης σε αυτό το σύστημα και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Αλλά όμως για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο μας νομίζω ότι προχωρούμε σωστά. Συνεργασία. Και υπάρχει εμάς αυτή η ατμόσφαιρα της συνεργασίας που κάτι που είναι ε, απαραίτητο. Κάτι κινείται. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε όλους και τους διερμηνείς. Όσους μας βοήθησαν. Και ελπίζω ότι η παρουσία σας εδώ θα βοηθήσει για να φτάσει εκεί που πρέπει το μήνυμα, να μας βοηθήσετε να φτάσει παντού το μήνυμα ότι υπάρχει και θα ισχύει αυτός ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και ελευθερίας.